Καλημέρα σε όλους. Yeah, guten Morgen. Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Δεν έχει ζητήσει κανείς κάποια αλλαγή υπήρχε αίτημα κάποιων συναδέλφων, εάν υπάρχει αίτημα κάποιων συναδέλφων να πάνε σε άλλες επιτροπές να... Επειδή κάποιοι συνάδελφοι να πάνε σε άλλες επιτροπές να ψηφίσουν, θα ψηφίσουμε αμέσως στις 9. Θεωρώ ότι αυτό εγκρίνεται. Δεύτερο ζήτημα τώρα, το γλωσσικό και Βεβαίως ευχαριστούμε την ε, διερμηνία και ούτως ή άλλως είναι δημόσια συνεδρίασή μας, μεταδίδεται στο ίντερνετ, οπότε θα ψηφίσουμε και ηλεκτρονικά σήμερα, οπότε σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες. Κύριε Γκάιερ, εγώ ακόμη δεν την ε, έχω την κάρτα μου, οπότε παρακαλώ για λίγα λεπτά να μπορώ να ψηφίζω με το χέρι. Μάλιστα. Οπότε ίσως μέχρι να περάσουμε, να ολοκληρώσουμε τα επόμενα σημεία της διαδικασίας, να έχει έρθει η κάρτα σας. Επί τη ευκαιρία συγχαίρω τον κύριο Ταβέν για τον ορισμό του στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εσωτερικό ελεγκτής, μάλιστα. Συγχαρητήρια και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για εσάς. Ja. Äh, Οπότε, λείπει σε κάποιον άλλον η κάρτα της ε, ψηφοφορίας. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε πρώτα απ' όλα μια δοκιμή. Μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχουμε ψηφοφορία. Ψηφίστε. Okay. Ένας από το ΕΛΚ είναι παραπάνω. Πέρας. Πέρας της ε, ψηφοφορίας όπως τα βλέπουμε εμείς από εδώ πέρα, είναι κάποιος παραπάνω από το ΕΛΚ. Έτσι είναι. Ωραία, ευχαριστώ. Άλλη μια δοκιμαστική ψηφοφορία, δεύτερη. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Äh, Πριν ε, περάσουμε στην ε, ψηφοφορία, θα ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ψηφίζουμε σήμερα μια σημαντική γνωμοδότηση. Δεν είμαστε εμείς η κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή. Την ε, βεβαίως η επιτροπή ε, νομικών θεμάτων γιατί ήρθαν σε εμάς διάφορα θεσμικά όργανα και μας τόνισαν τη σημασία αυτού του φακέλου. Θα ήθελα λοιπόν ε, εισαγωγικά ως πρόεδρος της Επιτροπής Ενέκτου Προλογισμού να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θεωρώ πως όλοι θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και βεβαίως το Κοινοβούλιο και η διοίκηση του Κοινοβουλίου και στο μέλλον να έχουν εξαιρετικό προσωπικό το οποίο βεβαίως θα έχει τα απαραίτητα προσόντα και θα εργάζεται με τον ανάλογο τρόπο για να μας βοηθήσει σε μια ορθή διοίκηση και καλή ε, νομοθεσία, καλή νομοθετική διαδικασία. Θεωρώ πως συμφωνούμε όλοι σε αυτά και θεωρώ πως ε, βεβαίως ε, αυτό είναι το βασικό μέλημα όλων των συναδέλφων. Το δεύτερο βεβαίως, το οποίο αναγκαία πρέπει να έχουμε κατά νου ως Επιτροπή Ελέγχου του Υπεροπολογισμού, είναι τα δημόσια οικονομικά. Τα δημόσια οικονομικά, τα λεφτά δηλαδή των φορολογουμένων κατ' ουσίαν, ε, λόγω κάποιας δύσκολης κατάστασης ε, σε κάποια κράτη-μέλη που, έχουν που έχει οδηγήσει σε κάποια δραστικά ε, μέσα λιτότητας ε, και στο σύμφωνο σταθερότητας ε, το οποίο βεβαίω αναγκαστήκαμε να υιοθετήσουμε για να προστατεύσουμε το κοινό μας νόμισμα αν σκεφτούμε το τι έγινε και στην Ουγγαρία, στη Λετωνία που είχαμε σοβαρές περικοπές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αλλά και στις δομές της αμοιβή στον δημόσιο τομέα Οπότε στο πλαίσιο αυτό κινούνται και οι τροπολογίες και δεδομένης της ε, σημασίας ε, ε, έλαβα μια ειδοποίηση πως η Κομισιόν θα ήθελε σε τρία λεπτά να τοποθετηθεί και ευχαρίστως βεβαίως να ανταποκριθώ σε αυτό το αίτημα. Οπότε τώρα θα δώσω τον λόγο στον κύριο Λαβασέρ από την Κομισιόν. Κύριε Λαβασέρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο. Τρία σημεία όσον αφορά την πρόταση που συζητάτε σήμερα. Το πρώτο, το πλαίσιο. Λίγη μέθοδος προσαρμογής ε, των αμοιβών των υπαλλήλων και άλλων ε, προσωρινών υπαλλήλων που λύγει 31 Δεκάτου 2012. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει οπωσδήποτε να λάβει πρωτοβουλία το δεύτερο είναι η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δίτη. Πρώτα απ' όλα να διορθώσουμε τις ανεπάρκειες που διαπιστώσαμε στην προηγούμενη μέθοδο, κάτι διάρκεια της εφαρμογής της και δεύτερη να υπάρξουν ουσιαστικές εξοικονομήσεις για την Ευρωπαϊκή Δημοσιοδίκηση διατηρώντας ωστόσο την ελκυστικότητά της για να απαντήσουμε λοιπόν και στο πλαίσιο και στη φιλοδοξία, η Επιτροπή προτείνει δύο μεθόδους, δύο δηλαδή μέτρα. Το πρώτο να μειωθεί ο αριθμός των υπαλλήλων στο σύνολο των ευρωπαϊκών οργάνων κατά 5% τα επόμενα 5 έτη και δεύτερο να τροποποιηθεί ο κανονισμός δημοσιοπολιτικής καταστάσεως. Βεβαίω περιορισμένα, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις σταδιοδρομίες. Στόχο επίσης όμως έχουμε και άλλα στοιχεία περιορισμένα ούτω ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα τη ε, Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκησης. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια μεταρρύθμιση όπως ε, την είδαμε το 2004, αλλά για μια αναθεώρηση και για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της λήξης ισχύω της μεθόδου και για να λάβουμε υπόψη την οικονομική κατάσταση στα κρατημέλη. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Λεβασέ. Δεν συνηθίζεται πριν από την, κομισιο... πριν από την συζήτηση να γίνει, πριν από την ψηφοφορία με συγχωρείτε να γίνει συζήτηση. Die ε, Γι' αυτό θα ήθελε τώρα να μιλήσει και η, η Εάν το επιθυμείτε να γίνει ε, ένας γύρος παρεμβάσεων, ε, ένα λεπτό ανά ομάδα. Αλλά εγώ προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Κύριε Οντή, συμφωνείτε? Να περάσουμε κατευθείαν στην ε, ψηφοφορία. Οπωσδήποτε θέλετε να μιλήσετε. Ωραία, ας ακούσουμε πρώτα την εισηγήτρια. Όχι, όχι, δεν θέλει. Ο κύριος Οντή. Θα ήθελα η Επιτροπή να διευκρινίσει ποια είναι η ποια είναι η φύση του κοινωνικού διαλόγου που έλαβε η χώρα για αυτήν ε, την πρόταση. Ο κοινωνικό διάλογο στα κράτη-μέλη είναι πολύ διαφορετικό. Πώ έγιναν τα πράγματα με του εκπροσώπου του προσωπικού, πώ διεξήχθη ο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα κύριε Λαβάσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Επιτροπή υπάρχει ένα σύνολο κανόνων σε σχέση με τον κοινωνικό διάλογο που γίνεται με τις ε, οργανώσεις που εκπροσωπούν το προσωπικό. Η Επιτροπή υπέβαλε το σχέδιο πρότασης στους εκπροσώπους του προσωπικού και το σχέδιο αυτό συζητήθηκε με τους εκπροσώπους του προσωπικού όλο το φθινόπωρο σε διάφορα επίπεδο, επίπεδα και σε τεχνικό, διοικητικό αλλά και πολιτικό επίπεδο με τον αντιπρόεδρο του προσωπικού ή επαγγελματικές ενώσεις ενημερώθηκαν, υπήρξε διαβούλευση καθ' όλη τη διάρκεια της ε, περίοδου που προηγήθηκε της υποβολή της πρότασης τον Δεκέμβριο. Ευχαριστώ. Νομίζω ξεκαθάρισε έτσι και ένα σημαντικό ζήτημα και περνάμε στην ψηφοφορία. Yeah, okay. Äh, ich schlage vor, dass... Προτείνω να ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί ίσως να είναι τσίμα τσίμα τα πράγματα. Άρθρο 1, παράγραφος 1, τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ωραία. Ξεκάθαρο. Άρθρο 1, άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, ε, τροπολογία 32. Ψήφισαν όλοι πέρας. Μάλιστα. Τροπολογία 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Και πέρας. Μάλιστα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. Έχει αλλάξει ελαφρώς η συμβαστική τροπολογία. Σα την μοίρασαν χθε το βράδυ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Όχι. Περνάμε στην ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβιβαστική Β. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Πρέπει λοιπόν τώρα να ψηφίσουμε χωριστά. 37. Σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο, άρχιτη ψηφοφορία. Για το πρώτο μέρος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Πέρας της ε, ψηφοφορίας. Δεκτή. Όχι, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται, σαφώς. Ναι, με συγχωρείτε. 35 καταπίπτει. 36. Καταπίπτει. Α, καταπίπτει. 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 39. 39. εννέα, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 41. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 40 την αποσύρει η συγγήτρια. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α και εδώ πέρα υπάρχει αλλαγή. Έχετε όλο το νέο κείμενο. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της α. α άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Και περνάμε με την προφορική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 55 σε δύο μέρη, σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο. Άρχη τη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Μέρος τρίτο. Άρχη τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Προσπερνάμε την 56 και περνάμε στην τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Κατόπιν 58 άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 59 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τώρα υπαρθμόν 60 σε δύο μέρη. Άρχεται η ψηφοφορία για το πρώτο μέρος. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Now we vote an amendment number one. Τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Unblock. Τροπολογίες 63 και 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Προφορική τροπολογία 2. Περιφορική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 64. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, δεκτή. 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Τοπολογία 2. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Τροπολογία 3. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Υπαριθμών 66. Όχι, καταπίπτει. Οπότε περνάμε στην τροπολογία 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 68. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι ακόμα. Πέρας. Δεκτή. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 70 καταπίπτει, 4 καταπίπτει. Περνάμε λοιπόν στην 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 72. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. 5 με συγχωρείτε. Άρχεται η ψηφοφορία. 5. Πέρας δεκτή. 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Ε, block... Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες μαζί τις ε, τροπολογίες 76 έως 79. Έχει κάποιο αντίρρηση. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε μαζί τις 76 έως 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία 80 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 80, 80. 8-0. την υπαριθμόν 80 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Η 6 καταπίπτει. Τροπολογία 81. Άρχεται τη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 82. Όχι, κα... ψηφίζουμε τον 82 μάλιστα. 82 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. 83. Πρέπει να ψηφίσουμε την 83, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας. It is taken. Εγκρίνεται. 84. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 85. Άρχεται. 85 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 86. Άρχεται 86. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 87. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 88. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 89. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 90. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 91. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Από κοινού. 5 και 6. Άρχεται. 5 και 6 από κοινού άρχεται. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 94. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 11. Καταπίπτει. 95. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 96. Να ψηφίσουμε μαζί 96-99. Έχει κανείς αντίρρηση. Ωραία, από κοινού. Ψηφίζουμε λοιπόν 96 έως 99 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λίγοι. Απορρίπτονται. Τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγοι. Απορρίπτονται. Τροπολογία 101. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. 102. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 103. Άρχεται. 103. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Άρχεται. Επί τις 12. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Ε, μία ψήφο. Πλειοψηφία. 13. Άρχεται. 13 λοιπόν. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. <coughs> Απορρίπτεται. 14. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Τροπολογία 15. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Από κοινού 16-18 άρχεται λίγη απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Οι 17 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απορρίπτεται. 19. Άρχεται. Λίγοι. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. Τροπολογία 20. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Λίγοι. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 24. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απορρίπτεται. 26. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι λίγοι. Εγκρίνεται. 27. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απορρίπτεται. 29. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Απορρίπτεται. 30. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Λίγοι. Εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της ε, γνωμοδότησης ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Λίγοι. Εγκρίνεται. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Την πολύ έντονη προετοιμασία και την ε, ψηφοφορία. Συγχαίρω την εισηγήτρια. Ένα σύντομο διάλειμμα, μια σύντομη διακοπή πριν συνεχίσουμε τις συνεδρίες. liebe Kolleginnen, Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε πολλή δουλειά. Πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ όσους θέλουν ε, να συζητήσουν μεταξύ τους, να ε, βγουν έξω. Συνεχίζουμε την ημέρη διάταξη. Δεν καλωσόρισα και να καλωσορίσω τώρα τον νέο συνάδελφο που διαδέχεται τον κύριο Ήτελε που πήγε στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο Χαιρετίζω τον, τον συνάδελφο Σάρβαμα Τελετούλουα στα φιλαδικά. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Ε, με συγχωρείτε ε, να πληρώσω, έπρεπε να το έχω κάνει προηγουμένως. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 4. Απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εισηγητής μας είναι ο Κρίστοφαρ Φιέλνερ που ανέλαβε την έκθεση από τον συνάδελφο Χάτζη Μαρκάκη στις 21 Φεβρουαρίου 2012. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε μια πρώτη έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 318 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση αυτή αφορά το 2010, την οικονομική χρήση 2010. Για τη σημερινή συζήτηση με μεγάλη χαρά Καλωσορίζω την Γενική Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Κάθριν Ντέι. Για άλλη μια φορά είναι παρούσα στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Και καταρχάς να σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ κυρία Ντέι και καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να εφαρμόσουμε το άρθρο 3.13 της συνθήκης. Η Επιτροπή σας ξέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να, να βελτιώσει τον τρόπο αξιολόγησης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε την ε, ε, αποτίμηση επιπτώσεων, εξάντε δηλαδή η εκτίμηση, Τώρα όμως θέλουμε και για τον ex αποτίμηση να κάνουμε περισσότερα. Θα διαπιστώσατε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία ελέγχου και εποπτείας στην πρότασή μας για το επόμενο πολιετές χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Οι αλλαγές αυτές φασίζονται κατά πολύ στην ανάλυση και αποτίμηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, να δούμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε και μερικά στοιχεία που αναφέρονται στην νέα πρόταση προέρχονται από τις αποτιμήσεις που προκύπτουν σε αυτήν την ε, αρχική έκθεση που σας υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η πρώτη έκθεση ανέδειξε πολλά ερωτήματα. Τι να καλύψουμε. Τι σχέση πρέπει να έχει με διάφορες άλλες ογκώδες εκθέσεις, άλλους ε, μηχανισμούς ε, λογοδοσίας και πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά με τη διαδικασία απαλλαγή. Όπως είπα, έχουμε την ετήσια έκθεση των γενικών διευθύνσεων, την συνθετική έκθεση που ε, εγκρίνει το Σώμα των Επιτρόπων θα θέλαμε λοιπόν να δούμε πώς θα κάνουμε στο μέλλον τις εκθέσεις αποτίμησης για να βοηθήσουμε τη δουλειά και τις επιτροπή σας. Η αποτίμηση φυσικά, η αξιολόγηση είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Δεν συνδέεται αυστηρά με τη διαδικασία απαλλαγής. Η απαλλαγή πολύ συχνά θα πρέπει να επικεντρωθεί σε θέματα για τα οποία δεν έχουμε τα αναγκαία στοιχεία από τη μισή. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πολλέ εκθέσει από μαζί, από κοινού, να εξετάσουμε πολλέ εκθέσει από κοινού για να συντονίσουμε την εργασία μα. Με βάση το άρθρο 318 λοιπόν, ακολουθήσαμε την ε, διατύπωση του άρθρου για να δούμε τι αποτελέσματα επέτυχαν τα προγράμματα τα οποία αποτιμούμε. Όπως ξέρετε, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό που είναι σημαντικά θέματα της Ευρώπης 2020 και που τα διαχειρίζεται απευθείας Επιτροπή σε πολλού τομεί. Και για αυτή τη συζήτηση σήμερα έχουμε πληροφορίε για τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα. Έχετε συνόψη των κυρίων στοιχείων μας. Θα δείτε ότι σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε ότι επέτυχαν τα προγράμματα αυτά, αλλά υπάρχουν βέβαια και τομεί βελτίωση. Θα πρέπει να έχουμε, για παράδειγμα, λέμε λιγότερου στόχου, να απλοποιήσουμε τη διαδικασία. Αυτά τα έχουμε ήδη συμπεριλάβει στι προτάσεις μας για το επόμενο πολιετέ χρηματοδοτικό πλαίσιο. Έχουμε καλύψει λοιπόν αυτού του τρει τομεί. και τώρα θα θέλαμε να καλύψουμε και άλλους τομεί ε, του χρόνου, για παράδειγμα περιφερειακή πολιτική, ενεργειακή πολιτική, μεταφορέ. και περαιτέρω το 2013, περαιτέρω άλλου τομεί δηλαδή, ούτω ώστε σε μερικά χρόνια να έχουμε καλύψει το πλήρε φάσμα των πολιτικών. Και κάθε χρόνο θα βασιζόμαστε και, τα στοιχεία, και στα στοιχεία που έχουμε για την πραγματική απόδοση. Αλλά θέλουμε να σας βοηθήσουμε με βάση τι είναι πιο χρήσιμο για σας. Έχουμε μια πρώτη έκθεση. Αναφέραμε μερικά από τα θέματα που εμάς μας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις σας και εφόσον έχουμε τις προφορίες εκ των υστέρων μπορούμε να δούμε και διαφορετικά τα θέματα, να τα παρουσιάσουμε διαφορετικά στην δεύτερη έκθεση που θα σας υποβάλουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος κυρία Ντέι. Να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον εισηγητή κύριο Φιέλνερ, αν το θέλει. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέη για την παρουσίαση της αξιολόγησης και της σχετικής έκθεσης Επιτροπής. Είχα γράψει στις σημειώσεις μου να την καλωσορίσω αλλά και αποσιοποιητικά. Τώρα θα περάσω κατευθείαν στα αλλά. Να σας πω ποιες είναι οι ανησυχίες μου. Πρώτον, ο κύριος ε, Μαρκάκη, εχθέ όταν μιλούσε για την απαλλαγή έριξε το βάρο σε αυτή την έκθεση αξιολόγηση και επί τη ουσία εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα από αυτέ τι 16 σελίδες ε, για να καλύψουμε τις απαιτήσει του άρθρου 313. Αλλά ίσως θέω εγώ, θα δω και πώς ε, αντιδρούν οι συνάδελφοι, αν είχα υπερβολικές προσδοκίε, δηλαδή. Αυτό που περιέπλεξε δε περισσότερο τη ζωή μου είναι τα περί όχι ότι έχουμε σχεδόν ε, τε, ολοκληρώσει, περατώσει τη διαδικασία απαλλαγής, έχουμε καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό και ως εκ τούτου είναι δύσκολο, όπως σωστά είπατε, να λάβουμε υπόψη την, ε, το πνεύμα ε, της πρότασης, ότι πρέπει να συνδυαστεί δηλαδή με την διαδικασία απαλλαγής. Είναι δύσκολο βεβαίως τον έχουμε καθυστερήσει τόσο να συντονίσουμε τις δύο διαδικασίες. Ε, ελπίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα καταθέσει τις παρατηρήσεις όπως υποσχέθηκε. Πιστεύω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και θα μας βοηθήσουν ε, στις προσπάθειές μας. Πάντως χρειαζόμαστε σε κάθε περίπτωση περισσότερο χρόνο και θα πρέπει να αποπειραθούμε να, να διαμορφώσουμε το χρονοδιάγραμμα με κάποιο τρόπο όταν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει αυτή την έκθεση αξιολόγησης. Ε, να πω κάτι διαφορετικό τώρα. Νομίζω ότι είναι θετικό που κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Αυτή η μεικτή διαχείριση, η κοινή διαχείριση, shared management, ε, δεν περιορίζεται σε αυτό που είπατε. Όταν προσπαθούμε να αποτιμήσουμε τις επιδόσεις, τα επιτεύγματα, γιατί βλέπουμε στην αξιολόγηση ότι είναι, δεν είναι ικανοποιητικά, ε, ικανοποιητικές επιδόσεις κάποιων κρατών μελών, και θα έπρεπε να δούμε με ποιο τρόπο σε όλη την αλυσίδα, καθ' όλη τη διαδικασία ε, διεξαγάγεται αυτή η αξιολόγηση. Με ποιο τρόπο επιθυμεί να αναβαθμίσει τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν ε, τρόποι, υπάρχουν διαδικασίες ε, βάσει των οποίων οι εθνικές αρμόδιες αρχές με κάποιον τρόπο θα μπορούσαν ε, να είναι υπεύθυνε για τον ε, συντονισμό των προσπαθειών Επιτροπής και κρατών μέλων για την κατάρρη τη έκθεσης Αξιολόγηση, Θα ήθελα μια απάντηση από αυτού. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω ε, κάτι που ήγηρε πέρσι ο κύριος Χατζημαρκάκης στη δική του έκθεση. Η ιδιοκτησία, δηλαδή τα πνευματικά δικαιώματα για την έκθεση. Εσείς είστε ο παραγωγός, αν θέλετε, της έκθεσης, μας την παρουσιάσατε όμως ο κύριος Χατζημιαρκάκης και όλοι εμείς ζητήσαμε να διοριστούν επί τούτο ε, άνθρωποι που θα ε, ε, είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή αυτής της έκθεσης και πάγια θα ασχολούνται με τη σύνταξη αυτών των εκθέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να δοθεί μια συνέχεια σε αυτή την περσινή συζήτηση. Επίσης, διαπιστώνω ότι δίνει... Ε, παρατηρείται καμία εξέλιξη του ρόλου των ε, μεσαζόντων κατά την αποτίμηση αυτών των ε, επιδόσεων. Ξέρω ότι δεν υπάρχει ηρμό στις ερωτήσεις μου, φύγω πολύ διαφορετικά ζητήματα αλλά πρώτη φορά συζητήτε το θέμα και είναι δύσκολο λοιπόν να ξέρει κάποιος τι μπορεί να περιμένει από μια τέτοια έκθεση. Ένα άλλο ερώτημα που με απασχολεί είναι το εξή. Το άρθρο 318 της συνθήκης μιλάει για τα αποτελέσματα, results, Πώς ορίζεται το αποτέλεσμα. Δεν έχω μεταφυσικές ανησυχίες. Ήθελα μόνο να ε, ε, καταλάβω πώς γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στην έκβαση και στο αποτέλεσμα. Outcome και result. Εγώ βλέπω ε, την έκβαση των προγραμμάτων, αλλά αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτόματα ως συγκεκριμένο αποτέλεσμα διότι δεν συνδέεται με δείκτες επιδόσεων Φερρυπίν Με στην έκθεση περιγράφεται, περιγράφονται η ιδού η έκβαση της όλης διαδικασία. Έτσι παρουσιάζεται το θέμα. Καλό θα ήταν όμω να αποφασίσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτήν ακριβώς ε, την διάκριση ανάμεσα στην γενική έννοια του, της έκβασης και του συγκεκριμένου αποτελέσματος. Θα σταματήσω εδώ για να ακούσω και τους συναδέλφους. Πάντως, ε, συνοψίζοντας, ε, θα επαναλάβω ότι ήταν δύσκολο να γίνει αυτό λόγω του χρονικού περιορισμού και δεύτερον, περίμενα περισσότερα πράγματα από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, απηχώντας και τις απαιτήσεις του άρθρου 318 της Συνθήκης. Ε, Ευχαριστώ κύριε Φιέλνερ. Ο κύριος Χατζημαρκάκης τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Ντέι. Καταρχάς ε, θα είμαι ευγενικός μαζί σας. Γιατί δεν είναι όλα πολύ ευγενικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βεβαίως Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή συνεργασία. Το ανέφερε ο εισηγητής για την πολύ καλή συνεργασία πέρυσι η οποία προκάλεσε υψηλέ προσδοκίε. Ε, συγκεκριμένα σε ένα σημείο. Ένα σημείο που είναι πολύ σημαντικό για το φορολογούμενο. Πάντα ελέγξαμε μέχρι τώρα την ε, νομιμότητα και κανονικότητα. Εμεί το ελεγκτικό συνέδριο όλων των δαπανών, εσεί για τον εαυτό σα. Και γενικά είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά την αποτελεσματικότητα, την επίπτωση με την έννοια αυτών που κάνουμε δεν έχουμε ασχοληθεί. Αλλά οι συνθήκε μα επιβάλλουν να ασχοληθούμε και με αυτό. Εσείς ε, επιμένετε στη διατύπωση του άρθρου, αλλά αγαπητή κυρία Ντέι, αγαπητή Επιτροπή, δεν αρκεί η διατύπωση. Δεν ε, δικαιώνουμε τον φορολογούμενο αν μετά από τόσα χρόνια ύπαρξη της Ένωσης δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε τι ακριβώς κάνουμε. Ο εισηγητής έχει δικαίωμα να μάθει τι κάνουμε τα λεφτά του, πώς τα διαχειριζόμαστε. Φυσικά υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Η έκθεση αποτίμησης είναι απλώς ένα όργανο του ε, δασκάλου προς τον εαυτό του. Δηλαδή απλώς ο μάνατζερ αποτιμά τι έχει κάνει. Θα έπρεπε λοιπόν να συνεργαστούμε περισσότερο. Στο τέλος θα κάνω μια πρόταση. Ξέρετε ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι διατεθειμένο να ελέγξει αυτή την έκθεση αποτίμηση και εκείνο. Να δώσει και αυτό με έναν τρόπο την απαλλαγή του. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξηγήσουμε στον φορολογούμενο. Σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά. Υποβλήθηκε λίγο καθυστερημένα αυτή η έκθεση. Είχα μεγάλε προσδοκίε, το ομολογώ. Περίμενα κάτι του ουσιαστικό. Γιατί το είχαμε συζητήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι που δεν θα το περίμενε κανεί. Αλλά όδιναν όρο και έτεκε μην. Σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Είμαι πολύ απογοητευμένο. Ιδιαίτερα γιατί συζητήσαμε προηγουμένω για τον κανονισμό ε, δημοσιο, δημοσιοϊπαλληλική καταστάσεω. Ε, σπάσαμε το κεφάλι μα, ψηφίσαμε και το, και το Κοινοβούλιο συνολικά φυσικά υποστηρίζει την Κομισιόν στι μεγάλε γραμμέ, στι γενικέ γραμμέ. Θέλουμε να έχετε επαρκέ και καλό προσωπικό. Αλλά αυτό το προσωπικό να μα τα παρουσιάζει έτσι τα πράγματα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θα μπορούσατε να τα έχετε πάει καλύτερα. Λέτε, εμείς βασιζόμαστε στη διατύπωση, διατύπωση του άρθρου. Έχουμε μια έκθεση 16 σελίδων. Αλλά δεν αναφέρεται τίποτα συγκεκριμένο σε 16 σελίδες. Πού έγιναν θέσεις εργασίας, δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, πόσες. Μόνο γενικές επιπτώσεις έχετε περιγράψει. Αυτό θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και μόνοι μας. Και πολλούς σημαντικούς τομείς δεν τους αναφέρατε. Ασχοληθήκατε με εκπαίδευση, έρευνα, πολιτισμό. Εσείς τους διαχειρίζεστε, καλά τα πάνε, αλλά δεν δαπανώνται εδώ οι περισσότερες δαπάνες. Υπάρχει μια λέξη στα γερμανικά, μια έκφραση στα γερμανικά, μπλα μπλα μπλα. Είναι απολύτως ασαφή αυτά. Δεν είναι, δεν αρμόζει στην Κομισιόν αυτό το οποίο έχει υποβληθεί εδώ. Το ανέφερε ήδη ο Φιέλνερ. Πέρυσι δώσαμε συγκεκριμένε κατευθύνσει. Τι θέλουμε. Θέλουμε για παράδειγμα δίκτες ε, αποτελεσματικότητας κλειδιά. Θέλουμε να συνδυάσουμε, να συγκρίνουμε του στόχους με το αποτέλεσμα. Εσείς τα είχατε συζητήσει, είχατε πει ότι συμφωνείτε και δεν βλέπω να αντικατοπτρίζονται εδώ στην έκθεση. Αγαπητή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν έπρεπε να αποφασίσω αν θα περάσετε τη χρονιά, θα αποφάσιζα ότι έχετε μείνει στην ίδια τάξη. Είμαι πολύ απογοητευμένος. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας εμείς για αυτή την αποτίμηση, για την έκθεση αποτίμησης. Έχουμε αρκετή πείρα και στην συνεργασία με το Ελεκτικό συνέδριο για να μπορέσουμε να εκπονήσουμε κατευθυντήρες γραμμές για εκθέσεις αποτίμησης στο μέλλον που να είναι πολύ διαφορετικές στο μέλλον. Βεβαίως μπορεί να ανταποκρίνονται οι εκθέσεις αυτές στο γράμμα, αλλά δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Ο, ε, ως Πρόεδρος δεν πρόκειται να κάνω πολιτικά σχόλια, αλλά διάβασα από την έκφραση των προσώπων των μελών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι εδώ των υπαλλήλων ότι είναι πολύ χαρούμενοι που δεν είστε δάσκαλό του και δεν αποφασίζετε αν θα περάσουν την τάξη. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ντέι, γνωρίζετε πως... Θα το πω. Εδώ, εδώ είμαι. Ξέρετε πως ε, βεβαίως ε, Έχουμε κάποια συμπάθεια για εσάς και για τη δουλειά σας, αλλά ε, αυτά τα οποία ακούσαμε από τους συναδέλφους βεβαίω ήταν μια σειρά παραπώνων και δυστυχώς θα πρέπει και εγώ να τα συνεχίσω γιατί αυτά τα οποία είπαν ε, ο κύριος Φιέλνε και ο κύριος Χατζημαρχάκης ε, δείχνουν κάποια πράγματα. Μιλάμε για ποιότητα και όχι ποσότητα, αλλά αν δούμε τις εκθέσεις του 2009 και ε, παλαιότερες. Οι αξιολογήσεις αυτές αφορούσαν όλους τους ε, τομείς ε, της πολιτικής. Ήταν πάρα πολλά χαρτιά, 169 σελίδες το 2008, 300 τόσες το 2009. Δεν λέω να μας στέλνετε τέτοια πάκα, αλλά σε σύγκριση με τις 16 σελίδες που μας στείλατε τώρα, ε, είναι μεγάλη η διαφορά. Και το είπαν νομίζω και οι δύο προλαλήσαντες. Ε, Βεβαίω, εντάξει, βεβαίως είπατε και εσείς πως πρόκειται μόνο για μία αναφορά για την ε, έρευνα, την εκπαίδευση, για λίγους ε, τομείς πολιτικής και λέτε του χρόνου ναι θα δούμε κάποιους άλλους τομείς της πολιτικής και σε μία περίοδο κάποιων ετών θα εξετάσουμε το σύνολο. Δεν νομίζω πως ήταν αυτό το νόημα όμως της ερώτησής μας. Ναι βεβαίως να έχουμε ε, μια καλή έκθεση της αξιολόγησης, αλλά βεβαίως η συνθήκη της Λισαβόνας έχει φροντίσει και το άρθρο 318 συγκεκριμένα να έχουν ένα κάποιο επίπεδο αυτές οι εκθέσεις. Δηλαδή, εντάξει, ασχολούνται μόνο με λίγους τομείς πολιτικής για ακριβώς για να είναι πιο ποιοτικές ε, και το είπε και ο κύριος Χατζημαρκάκης. Κατόπιν έχουμε το χρόνο, το είπε ο κύριος Χέλνερ. Οι προηγούμενες εκθέσεις αξιολόγησης ήταν διαθέσιμες ε, τον Μάιο του επομένου έτους ε, του οικονομικού. Τώρα τις ε, έχουμε εννέα μήνες αργότερα. Δηλαδή ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Το είπε και ο κ. Χελνέρ, δεν δυσκολεύει έτσι η δουλειά μα. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε την απογοήτευσή μα και τι ε, παρατηρήσει μα τι επικριτικέ. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια παρεξήγηση δηλαδή. Ε, δηλαδή μας λέτε επισήμω, ναι, σύμφωνα με το άρθρο 318 ε, και αυτά τα οποία αναφέρει τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Έχουμε μία έκθεση αξιολόγηση. ναι το δέχομαι, αλλά Πού είναι η αρχική αξιολόγηση που είχαμε, που ήταν πολύ περισσότερα πράγματα. Αν μας το εξηγήσετε αυτό, θα είμαστε ικανοποιημένοι. Ναι, σας ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα τον ε, Γιάν Μούλτερ σε αυτό το κύριο ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή Για πρώτη φορά αυτή η έκθεση δείχνει μείωση των ε, επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι λυπηρό. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν έρθει αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα για 17 ε, συναπτά έτη. Είναι αρνητικά ε, τα αποτελέσματα, δεν υπάρχουν θετικά στοιχεία και το θέμα είναι με ποιο τρόπο πρέπει να αντιδράσουμε στο παρελθόν. Ω επιτοπλίστων σας έδωσε μια ευκαιρία το Κοινοβούλιο με την απαλλαγή. Αμφιβάλλω αν θα συμβεί αυτό φέτος. Διότι αυτή τη χρονιά όπου η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα ελλημάτων, Κάποιοι έχουν θετικέ επιδόσει, αλλά τέλο πάντων όχι η πλειοψηφία. Απευθύνονται επικρίσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση του προπολογισμού και συνειδητοποιούμε ότι δεν δύναται να λάβει την δήλωση αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ελεγκτικό ε, συνέδριο. Μειώνοντα έτσι τις δαπάνες, τις κρατικές δαπάνες όλων των κρατών μελών τη ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ δύσκολα μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό στο κοινό. Για ποιο λόγο δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα μετά από τόσα χρόνια να ε, ε, επιτύχετε αυτές τις θετικέ επιδόσεις που περιμένουμε. Ε, το Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι βάσει της διαθεσμικής, διοργανικής μάλλον συμφωνίας ε, προβλέπεται πλέον κάτι που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο, οι αιτήσιε ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις. Ε, η συμφωνία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει αιτησίως να υποβάλουν εκθέσεις και για ποιο λόγο το ζητήσαμε, ώστε να μπορέσουν να νιώσουν πιο υπεύθυνα τα κράτη-μέλη σχετικά με τη διαχείριση των κονδυλίων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία, παράγονται πλέον αυτές οι αιτήσει εκθέσεις. Πλην όμω ε, είναι μυστικέ και το δεύτερο μέρο τη συμφωνία ε, διαβαθμίζει αυτέ τι εκθέσει. Πόσο γελίο είναι αυτό. Τα τρία θεσμικά όργανα κάνουν μια συμφωνία, εκτελείται η συμφωνία, όμω με τη συγκατάθεση τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή αναφέρεται ότι ε, τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν έχουν πρόσβαση, σε, ή μάλλον τα θεσμικά όργανα δεν έχουν πρόσβαση πέραν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτέ τι εκθέσει ε, των κρατών μελών. Για ποιο λόγο μπορείτε να μα εξηγήσετε, κρίνετε ότι είναι σωστά αυτά που κάνετε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κύριε Αντέι να σας δώσω την ευκαιρία να απαντήσετε συνολικά στις ερωτήσεις. Όπως τα καταλάβατε, η Επιτροπή, ανεξάρτητα από πολιτικές ομάδες, ε, είχε μεγάλες προσδοκίες ε, από αυτή την έκθεση αξιολόγησης και έχει ακόμη και περαιτέρω ερωτήσεις. Ίσως θα μπορούσατε παρακαλώ να μας δώσετε μερικές απαντήσεις που να μας δώσουν κάποια ελπίδα για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα αρχίζοντας ε, να δεχτώ την πρόσκλησή του κυρίου Στάζη. Όντως υπάρχει παρανόηση. Κατά τη γνώμη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έκθεση που προβλέπεται στο 318 είναι επιπρόσθετη σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε. Δηλαδή, συνεχίζουμε όπω και στο παρελθόν να δημοσιεύουμε και να κοινοποιούμε τι εκθέσει μα. Ε, και ε, πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα. Δεν κρίναμε ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα συμπίλημα όλων των εκθέσεων μέσα σε αυτή την έκθεση. Θα ήταν αδύνατο αυτό. Ε, αλλά θέλαμε να προσθέσουμε κάτι στη συζήτηση, δηλαδή προσθέτω πέραν από όλα αυτά που κάνουμε στα πλαίσια τη διαδικασία αξιολόγηση, χρειαζόμασταν κάτι για να κάνουμε ένα παραπάνω βήμα. Ε, και ρίχνοντα το φω σε κάποιου τομείς ανά έτος, θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να του αναδείξουμε σε ε, προτεραιότητα. Ούτω ή άλλω όλα τα υπόλοιπα διαδικτυακά και γραπτός δημοσιεύονται, κοινοποιούνται, είναι διαθέσιμα, αν θέλετε κάτι πιο λεπτομέρε. Αν λοιπόν θέλετε κάτι, ε, τι να σας πω, περιεκτικό όπως μια εγκυκλοπαίδεια, να την κάνουμε. Αλλά δεν ερμηνεύουμε εμείς έτσι ε, τη διατύπωση του άρθρου 318 και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, γίνει ένας εσωτερικός διάλογος. Δηλαδή, τι θα συντάξουμε θα σας βοηθούσε εσάς. Το συμπίλημα δεν ωφελεί αν δεν χρησιμοποιηθεί, αν δεν σας φαίνεται εσάς χρήσιμο. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι ο τρόπο, η μέθοδο που ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση. Πέρυσι, θυμάμαι, ήμασταν εδώ και συζητούσαμε την έκθεση του κ. Χατζημαρκάκη και ε, πιο συγκεκριμένα για τα διαρθρωτικά ταμεία λέγαμε ότι θέλουμε να ε, ε, προσανατολιστούμε προ τα αποτελέσματα και όχι προ τα δικαιώματα των περιοχών. Γι' αυτό και έγιναν σχετικέ προτάσει στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, τέλος πάντων είναι πάρα πολύ δύσκολες συζητήσει με τα κράτη-μέλη για αυτό το θέμα. Πάντως προσπαθήσαμε τα ταμεία ε, να ε, συνδεθούν με τις υποκείμενες ε, προτεραιότητες και προσπαθήσαμε τα κράτη-μέλη να είναι υπεύθυνα να μα καταδείξουν με τα αποτελέσματα να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και ελπίζω ότι θα έχουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για αυτή τη διάσταση της πρότασής μας, δηλαδή να ορίσουμε ποιο είναι ο στόχο η χρήση αυτών των κονδυλίων και κατόπιν αναφορά των αποτελεσμάτων. Δεν έχουμε φτάσει εκεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πάντω, συντάξαμε αυτέ ε, τι ε, προτάσει επί τη βάση των αξιολογήσεων και σα παραπέμπω σε αυτή την έκθεση που σα διαβιβάσαμε. Βλέπετε με ευκρίνεια την αρχιτεκτονική του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, διότι αναφέρθηκε ότι είχαμε πολλέ κατακαιρματισμένε όμω ε, δυνατότητε παρέμβαση και χρηματοδότηση, οπότε είναι δύσκολο με λογικό και χρήσιμο χρήσιμο τρόπο στη συνέχεια να υποβάλουμε εκθέσει επιδόσεων, να δούμε τι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Στη συνέχεια ε, κάναμε τη σύνδεση με τι ε, ανακράτο ε, σύσταση βάσει των νέων διαχειριστικών μεθόδων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διαρθρωτικά ταμεία και προσπαθήσαμε στη συνέχεια να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τα αποτελέσματα. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα συμφωνήσουμε επί των αδρών γραμμών και με την πάροδο των ετών, με την εφαρμογή του νέου συστήματο, ελπίζω να μπορέσουμε τελικά να επιτύχουμε με το στόχο μας. Ε, πάντως είναι προϊούσα η διαδικασία, δεν, είναι, δεν έχει ακόμη αποκρισταλωθεί. Τώρα, ε, για τα ειδικά σημεία, πρώτον για το χρονοδιάγραμμα, ε, Είπα ήδη ότι στα μέσα Νοεμβρίου θα υποβάλουμε την επόμενη έκθεση και ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα ως προς το χρονοδιάγραμμα για σας. Πάντως δεν θα μπορέσουμε, όχι επειδή δεν το θέλουμε, αλλά διότι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίε, δεν θα μπορέσουμε να συνδέσουμε ε, την κάλυψη της ετήσιας απαλλαγή με τα αποτελέσματα των επιδόσεων που θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη χρονική στιγμή. Το αναγνωρίζω κύριε Φιέλνερ ότι στο μέλλον θα έχουμε αυτό το πρόβλημα και όντω θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και είμαστε ανοιχτοί σε ε, συστάσει από πλευρά σα. Σίγουρα θα θέλαμε να εξετάσουμε το θέμα της κοινή διαχείρισης, shared management, είναι δύσκολο. Ε, δεν έχουμε την ευκταία συνεργασία ε, ως προς την προσκόμιση στατιστικών στοιχείων από πλευρά των κρατών μελών σχετικά με τις αιτήσεις εκθέσεις. 15 ε, τέτοιες εκθέσεις έχουμε υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έγκριση των κρατών μελών έχουν εγκριθεί αυτές οι εκθέσεις και έχουν διαβιβαστεί ε, στο Κοινοβουλίο ως προς την ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα. Σε κάθε γάμα δέλτα υπάρχει μονάδα αξιολόγηση σχεδόν σε όλες τις γενικές διευθύνσεις και αυτοί οι άνθρωποι ε, είναι αρμόδιοι για την ε, αξιολόγηση. Ήδη υπάρχει το σύστημα, κύριε Φιέλνερ, σε σχέση τώρα με το ρόλο τη Υπηρεσία Εσωτερικών Ελεκτών. Γνωρίζετε ότι είναι ανεξάρτητοι ελεγκτέ και άρα δεν μπορούμε να του επιβάλλουμε μέθοδο εργασία. Ε, Πάντω μα εξηγούν ποια μέθοδο χρησιμοποιούν και στη συνέχεια που δίνεται πιέζουμε ούτω ώστε να, πι... να βασίζεται η αξιολόγηση στι επιδόσει. Ο στόχο μα είναι η πολιτική να είναι κυκλική, δηλαδή πρωτού προχωρήσουμε μπορούμε να κοιτάζουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και να ε, ε, ε, βασιζόμαστε στο περιεχόμενο της έκθεσης αξιολόγησης κατά τον σχεδιασμό των επομένων πολιτικών. Τώρα, σε σχέση με μελλοντικά προγράμματα εργασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τα νέα σημεία κάνουμε την επαλήθευση αν υπάρχει έκθεση αξιολόγηση και αν έχει ληφθεί όντω υπόψη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε εν και δεν αναφέρονται μέσα σε αυτή την έκθεση και ξαναλέω, τονίζω, είναι επιπρόσθετη σε σχέση με άλλες δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η έκθεση. Αν θέλετε τώρα κάτι πιο γενικό, δεν ξέρω, θα σας βοηθήσει, θα είναι πιο γενικό και ούτως ή άλλως υπάρχουν αυτά τα δεδομένα σε άλλους τομείς. Κάναμε, εν πάση περιπτώσει, μια πρώτη απόπειρα για να προσθέσουμε, να προσφέρουμε και κάτι άλλο. Αν δεν σας βοηθάει όμως, αν ε, δεν ε, δημοσιεύονται παρκώς οι πληροφορίες ε, κατά την γνώμη σας, θα πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά πάντως εμεί έτσι βλέπουμε το θέμα αυτή τη έκθεση. Σα ευχαριστώ για το δεύτερο γύρο. Έχω ήδη 7 συναδέλφου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Σα παρακαλώ όλου να είστε σύντομοι. Ε, παρακαλώ. Um, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη, το νόημα της Ευρώπης και ολόκληρο το σκεπτικό δέχεται πίεση αυτή τη στιγμή λόγω της κρίσης του ευρώ, της οικονομικής κρίσης, λόγω του ότι κάποιες χώρες δεν θέλουν να πληρώνουν όσο πληρώνουν αυτή τη στιγμή και θεωρώ πως το όλο ζήτημα της προστιθέμενης αξίας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι ο βασικός τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η ευρωπαϊκή κρίση. Οπότε θεωρώ πως η αξιολόγηση της ε, πολιτικής μας είναι κρίσιμη. Εάν δεν μπορέσουμε να επιδείξουμε πως ε, όλα τα έργα τα οποία χρηματοδοτούμε με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν έχουν επαρκή προσθέμενη αξία, τότε έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα από ό,τι πριν. Γι' αυτό θεωρώ πως ειδικά τα θεσμικά όργανα όπως ε, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν υψηλότερη προσθέμενη αξία. Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής από το 2009 και με έχει εντυπωσιάσει το έργο του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά απογοητεύτηκα από τα αποτελέσματα πολλών πολιτικών μας. Αν δούμε συνολικά την ε, γεωργική πολιτική, τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα Εντό της αγροτικής πολιτικής. Ε, δεν πιστεύω αυτά τα οποία βλέπω το πόσο λιγότερα πράγματα επιτυγχάνουμε με τα τεράστια κονδύλια που έχουμε. Αν και συγκριτικά είναι μικρά. Σε απόλυτα νούμερα όμως είναι μεγάλα ποσά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πολύ πιο πολιτικό το ζήτημα. Εγώ θεωρώ πως ε, πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο στην αποτελεσματικότητα της ε, πολιτικής μας. Γι' αυτό πριν από δύο χρόνια ξεκίνησα να ζητάω από το ελεγκτικό συνέδριο στην ετήσια έκθεσή τους να μην κοιτάνε μόνο το πώς το ταξιδεύουμε αλλά και το τι επιτυχάνουμε. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τους ε, συναδέλφους που μίλησαν στον πρώτο γύρο και θα πω πως πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο πολιτικό βάρος στην αξιολόγηση της πολιτικής μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιάνν Μπάντι Να υπενθυμίσω πως η κυρία Μπέι μας είπε πως στις 10.30 πρέπει να φύγει. Απλά το υπενθυμίζω. Μπαλτσίτης κατόπιν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα εγώ να υπερασπιστώ την Κομισιόν. Πρόκειται για την ε, πρώτη έκθεση που εστιάζει σε συγκεκριμένους ε, τομείς ε, πολιτικής και βεβαίως οπότε δεν είναι εύκολο να συντάξει κανείς τέτοιες εκθέσεις και σας συγχαίρω για το ότι σήμερα έχουμε μια έκθεση η οποία μας δίνει μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει και μπορεί έτσι να προωθήσει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το τι μπορούμε να επιτύχουμε με τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά Βεβαίω ε, έχω και κάποιες ερωτήσεις. Το 2009 ο κύριος Μπαρόσο παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης και είπε πως η διαδικασία της Μπολόνιας δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά και πως το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και είμαστε πίσω από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, ακόμα και την Κίνα και πως χρειάζεται μία συνολική αναθεώρηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω Πώς πάμε, πώς προχωράμε. Η δήλωση αυτή έγινε πριν από δυόμιση χρόνια. Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον τομέα της ε, εκπαίδευσης και της ε, έρευνας. Και πότε νομίζετε πως θα επιτύχουμε αυτά τα οποία έθεσε ο κύριος Μπαρόσο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σαρβάμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, ε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ε, να πω κάτι ως νέος βουλευτής, γιατί ε, με κάθε σεβασμό σας μεταφέρω νέα από τον έξω κόσμο και θεωρώ πως το σημαντικότερο ζήτημα από αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα είναι το πως φαίνονται όλα αυτά προς τα έξω, προς τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους Φιέλνερ και Γερμπράντι και τον κύριο Χατζημαρκάκη. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν, αλλά θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Πρέπει να είναι λογικά αυτά τα οποία λέμε εδώ πέρα. Να βγάζουν κάποιο νόημα και αντιλαμβάνομαι οπωσδήποτε θα σας δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις και πρέπει να συνεργαστούμε αλλά όπως είπα το σημαντικότερο είναι ας πούμε στους πολίτες το τι πραγματικά αγοράζουν με τα λεφτά τους. Ε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Χατζημαρκάκης. Θα ήθελα να συμφωνήσω κυρία Ντεή με αυτό το οποίο είπατε για το Ταμείο συνοχή, πω πράγματι τώρα η Κομισιόν έχει στόχο αποτελέσματα. Και σα συγχαίρω, δεν πρέπει να ντρέπεστε. Γιατί δεν μα λέτε λοιπόν στην έκθεση αυτά τα πράγματα. Αυτό περιμένουμε. Δηλαδή αν λέτε πως θέλουμε, αν λέγατε θέλουμε να κάνουμε ένα διάλογο για να δούμε πώς θα δείτε τις ε, εκθέσεις μας. Ναι, τι άλλο θέλουμε ούτω ή άλλω υπάρχει ευρύτατη πλειοψηφία και είμαι σίγουρος πω όπως και η περσινή έτσι και η φετινή έκθεση θα σας δώσει κάποιες ε, κατευθύνσεις, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να ε, συντάξουμε μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που ακούω πως ε, στο μέλλον θα λαμβάνουμε την έκθεση τον Νοέμβριο. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το ότι δεν γίνεται αμέσως, αλλά πρέπει και εμείς να μπορούμε να κάνουμε την δουλειά μας. Και ο Νοέμβριος βέβαια είναι πολύ πιο πρακτικός από αυτό που έγινε φέτος. Ε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί δεν συζητάμε την ουσία, αλλά τη διαδικασία. Αλλά αυτό οφείλεται στο ότι ε, είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο θέλω να λάβετε υπόψη για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα, ε, δείκτες απόδοσης. Δεν υπάρχουν εδώ πέρα, εμάς μας αρέσουν. Δεύτερον, θεωρώ πως πρέπει να έχουμε μια σαφή περιγραφή της αρχικής κατάστασης. Μια βάση, με, βάση την οποία αξιολογούμε το εάν ε, οι δράσεις ήταν χρήσιμες ή όχι. Τρίτον, όλοι γνωρίζουμε πως είναι μακροπρόθεσμα τα προγράμματα και είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω πως πρέπει να ορίσουμε κάποιες ε, ενδιάμεσους και μετρήσιμους στόχους έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε το εάν έχουμε πορεία προς το τελικό αποτέλεσμα. Και τρίτον, η συνθήκη ε, μας υποχρεώνει να εστιάσουμε στα αποτελέσματα ε, τα οποία έχουν επιτευχθεί. Οπότε μια ανοιχτή διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να αποφεύγεται. Αυτά θα ήθελα λοιπόν να δείτε εσείς ε, για του χρόνου για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο εμείς θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ κύριε Φιέλνερ. Κυρία Ντέι, νιώθετε πως υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες ε, στην Επιτροπή μας από εσάς. Ο Χερμαν ε, Έσε, ο Γερμανός συγγραφέας, είχε γράψει πως κάθε αρχή κρύβεται ένα θαύμα και τα λοιπά. Ελπίζουμε λοιπόν αυτό το θαύμα να γίνει και στην διαδικασία αξιολόγησης, αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να μαγευτεί με θαύματα μια Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού, γιατί έχουμε συγκεκριμένες ε, ε, και βαθύτατες ε, προσδοκίες. Ακούμε παραδείγματος χάρη την Επιτροπή Προπολογισμού πως φοβούνται πως η απόφαση του Κοινοβουλίου ότι η Κομισιόν δεν θα δώσει ε, δεν θα δίνει κονδύλια για τηλεοπτική κάλυψη της ε, Κομισιόν δεν θα εφαρμοστεί. Όταν μιλάμε για αξιολόγηση και συγκεκριμένα αποτελέσματα, νομίζω καλό είναι να εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Μπορεί να φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά για εμάς δεν είναι. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε πως ε, στο μέλλον θα εφαρμόζονται αυτές οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Ίσως, νομίζω, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι σε ένα τελευταίο γύρο. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να ξεκινήσω με το τελευταίο σχόλιο περί προσθέμενης αξίας με το οποίο συμφωνώ. Νομίζω πως είδατε την ε, πολύ ουσιαστική έκθεση για την ε, προσθέμενη αξία που δημοσιεύσαμε μαζί με, το, με τις προτάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πρόγραμμα. Εκεί πέρα εξηγούμε στον πολίτη πού βρίσκεται η προσθέμενη αξία και είναι γεμάτη παραδείγματα με αριθμούς, με παραδείγματα του πώς έκανε τη διαφορά ε, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα μπορούσαμε να τα είχαμε επαναλάβει όλα αυτά σε αυτή την έκθεση, αλλά δεν βλέπω ποια θα ήταν αυτή η προσθέμενη αξία. Είχαμε την ε, ιδέα πως ε, οτιδήποτε κάνουμε εδώ πέρα είναι διαθέσιμο στην Επιτροπή σας και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι επιπλέον. Μπορούμε βεβαίως ε, να κάνουμε ξανά, όπως είπα, μια πλήρη παρουσίαση των όσων κάνουμε. Αν θέλετε αυτό θα κάνουμε. Αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι πιο καινοτόμο, μια, θέλετε, απόσταγμα των μακροσχελέστερων εκθέσεων αξιολόγησης που είναι διαθέσιμες Πράγματι κύριε Φιέλνερ ε, όλα αυτά τα ορόσημα υπάρχουν μέσα στην πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, οπότε όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί στις νέες προτάσεις. Αλλά οι νέες προτάσεις πρέπει να υιοθετηθούν, μετά να ξεκινήσουν τα προγράμματα και θα χρειαστεί λίγος χρόνος. Για το ερώτημα περί εκπαίδευσης. Έχουν συμβεί πολλά από όταν έκανε τη δήλωσή του το 2009 ο πρόεδρος, ο κ. Μπαρόζο, ειδικά όσον αφορά την προσέγγιση του 2020. Γιατί ξέρετε πως έχουμε ποσοτικούς στόχους, δύο από αυτούς ε, όσον αφορά την εκπαίδευση, ε, μία για όσους ε, φεύγουν χωρίς ε, τυπικά προσόντα από το σχολείο και μία για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σημειώνουμε την πρόοδο που κάνουμε κάθε χρόνο. Κάποια κράτη-μέλη πηγαίνουν καλά και υπερβαίνουν τους στόχους, κάποια άλλα όχι, οπότε εστιάζουμε μετά σε αυτούς οι οποίοι δεν πάνε όσο καλά θα ήθελαν και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Οπότε είμαστε σοβαροί άνθρωποι, ακούμε, κοιτάμε τους μηχανισμούς και δίνουμε κάποια συνέχεια. Αλλά δεν είναι τόσο ε, γρήγορη διαδικασία όσον αφορά τα αποτελέσματα, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε με τους δείκτες, πρέπει να τους εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, αλλά τώρα για δεύτερη συνεχή χρονιά μπορούμε να παρακολουθήσουμε το κάθε κράτος μέλος ε, ανάλογα με τους στόχους του. Οπότε βλέπουμε τώρα το που χρειάζεται που χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις. Αυτά θα πω μόνο κύριε Πρόεδρε, βεβαίως από τη συζήτηση αυτή και τα όσα ακούστηκαν, ακούμε ε, τα ποια είναι, ποιες είναι οι επιθυμίες σας. Αν μπορούμε να κάνουμε το χρόνου μια γενική σύνοψη, αν αυτό προτιμά η Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντέι για τις απαντήσεις σας, τη δυνατότητα που είχαμε να συζητήσουμε μαζί σας. Πιστεύω, αυτό που είπε και ο συνάδελφος Μπαλτσίτης, Ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη έκθεση αξιολόγηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε ήδη κάνει την προσφορά να μας δώσετε την ευκαιρία να σας δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αποτίμησης και προτύπων. Οπότε θα δούμε πώς εμείς θα εφαρμόσουμε την πρόταση αυτή που κάνετε για τα benchmark. Ευχαριστώ πολύ. Benchmark. Okay. Okay, the next, uh, Επόμενο θέμα στην μέση διάταξη. Ε, θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά από ό,τι έχετε τυπωθεί. Έχουμε την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και για τα δύο σημεία. Η συγκητής μα είναι ο συνάδελφος Ριβελίνη. Να συζητήσουμε λοιπόν και τι δύο εκθέσει. Για την ανταλλαγή λοιπόν απόψεων, καλώ πρώτα απ' όλα τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού συνεδρίου, καλωσορίζω τον κύριο Χάραλντ Νόακ, και του δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει το θέμα. Αξιότιμοι βουλευτέ, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Όπως σας είπα και τον περασμένο Δεκέμβρη, θέλησα να προετοιμάσω μία ειδική έκθεση και τώρα ολοκληρώσαμε την ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το 2012 για τα χρηματοοικονομικά μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ. Ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτήν την έκθεση για πρώτη φορά θα έλεγα θα δημοσιευθεί επίσημα η έκθεση την επόμενη εβδομάδα ε, κατά την ε, συνήθη διαδικασία. Πρώτα δημοσιεύουμε και στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνήθως, αλλά ε, δέχτηκα να κάνω το αντίστροφο για να επικοινωνήσει καλύτερα το ελεγκτικό συνέδριο με το αξιότιμο μέλη της Επιτροπής. Σας στείλαμε λοιπόν αντίγραφα εκ των προτέρων την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη Τρίτη είχα την δυνατότητα στο Στρασβούργο να κάνω ανταλλαγή απόψε με τον εισηγητή σας κύριο Ριβελίνη για τα κύρια σημεία και πορίσματα της έκθεσης. Η κυρία Φρόντινσάιν θα γυρνάει τις σελίδες, η βοηθός μου. Θα καλύψουμε τα εξή σημεία. Πρώτον, θα ορίσω τα χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Δεύτερον, θα παρουσιάσω τους κύριους λόγους για τι χρειάστηκε ένας τέτοιος έλεγχος. Θα περάσω στους κύριους στόχους, το εύρος και την προσέγγιση του ελέγχου και συνόψη των πορισμάτων και συστάσεων και φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στα σχόλια ερωτήσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα χρησιμοποιήσω μερικές, μερικά ακρονίμια αλλά έχετε στην έκθεσή μου ένα γλωσσάρι με όλες τις συντμήσεις και ακρονίμια αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι διαφορετικά από τις παραδοσιακές επιδοτήσεις. Στα πλαίσια του ε, πλαισίου μας έχουμε από τη μία συμμετοχικές συμμετοχές, εγγυήσεις και δάνεια που δίνουν δάνεια που πρέπει να αποπληρωθούν κατόπιν. Όταν επιστραφεί αυτή η χρηματοδότηση από τις ΜΜΕ, τότε μπορούν να ξαναχρηματοδοτηθούν, να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα μέχρι να λήξει το μέσο. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται, μπορεί να έχει αποτέλεσμα η δράση αυτού του μέσου εάν ε, χρησιμοποιηθεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαχείριση ε, των πόρων της συνοχής σημαίνει ότι τα μέσα αυτά χρειάζονται την ενεργό συμμετοχή των δημοσίων αλλά και ιδιωτικών ε, χρηματιστικών ιδρυμάτων. Τα ιδιωτικά λέγονται συνήθως τράπεζες. Τα, χρήματα, τα μέσα αυτά αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχουν στόχο να προσελκύσουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από ιδιωτικούς επενδυτές. Τέλος, όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, η πλειοψηφία των οργανισμών που χρησιμοποιούν τέτοια χρηματοοικονομικά μέσα διαρθρώνονται γύρω από ένα βασικό ταμείο holding fund, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια στο κέντρο. Ε, όμως αυτό είναι προαιρετικό. Η πολιτική συνοχή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ε, οικονομικής, ε, κοινωνικής και εδαφική συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντα τι διαφορές ανάμεσα στις επιμέρους περιοχές. Ε, γι' αυτό η βασική στόχη της πολιτικής είναι να επισπεύσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης επιλέξιμες για αυτά τα ταμεία περιοχές. Αναγνωρίζεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και αντιστοιχούν στο 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και άρα είναι κλειδί για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, την ευημερία και την, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόλησης. Δεν είναι νέα αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα, πάντως ε, αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Για την περίοδο 2007 2013, αυτή την προγραμματική περίοδο, περίπου 400 400 τέτοιοι οργανισμοί που χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά μέσα θεσπίστηκαν με πρικοδότηση άνω των 10 δις ευρώ. Όπως ε, βλέπετε στην πέμπτη έκθεση για την πολιτική συνοχή, προορίζεται να παίξουν, προορίζονται για έναν καταλητικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωσή της πολιτικής συνοχής μετά το 2013. Η τωρινή κρίση και η έλλειψη κεφαλαίων αυξάνει τις δυσκολίες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προς την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη χρηματοδότηση που χρειάζονται για τις δραστηριότητες τους. Επίσης, οι βασικοί φορείς, η Επιτροπή σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο καταδεικνύουν αυξανόμενο ενδιαφέρον σε σχέση με τις επιδόσεις αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων για την επίτευξη των στόχων τη πολιτικής και να αποφύγουμε εγγενεί κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα μέσα. Οι αρμόδιοι για την εκτέλεση διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους. Ο βασικός ε, στόχος του ελέγχου ήταν να αξιολογήσουμε τις δαπάνες του ΕΤΠΑ για τα χρηματοοικονομικά μέσα με αποδέκτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν αποτελεσματική η δράση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και γι' αυτό το λόγο εστιάσαμε την προσοχή μας σε τρεις βασικές πτυχές του ζητήματος. Πρώτον, ποιότητα της αξιολόγησης ε, των δανειακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, που κρίνει το βαθμό δημόσιας παρέμβασης στον τομέα. Δεύτερον, ε, αν το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΤΠΑ είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα και τρίτον η αποτελεσματικότητα των ίδιων των μέσων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Όσο πιο αποτελεσματικά είναι τα χρηματοοικονομικά αυτά μέσα, τόσο μεγεθύνεται η συνεισφορά τους στην ε, τόνωση της ανάπτυξης και στην αύξηση των θέσεων απασχόλησης ο εσωτερικός έλεγχος εκάλυψε την περίοδο 2000 2006 ε, και 2007 2013 και τις δύο προγραμματικές περίοδους. Λοιπόν, για την πρώτη ολοκληρώθηκαν όλα τα προγράμματα ε, και τα Υπάρχουν κάποια δε που πλησιάζουν στο τέρμα τους ε, για το 2007-2013. Μετά από την πενταετία ε, ε, τα μία αυτά θα έπρεπε να ακολουθήσουν την ε, φυσιολογική διαδικασία, να συνεχίσουν να τρέχουν δηλαδή τα προγράμματα που είχαν ήδη ξεκινήσει, εντοπίζοντας βασικοί παίκτες και η Επιτροπή και τα κρατημέλη για τη χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων και κυρίως σε επίπεδο κράτους μέλους. Ένα δείγμα 34 επιχειρήσεων τιτλοποίησης και έκδοσης δανείου σε πέντε κράτη-μέλη εξετάστηκαν, σχεδόν δηλαδή 40% των των δεσμεύσεων, των δεσμευμένων κονδυλίων για την περίοδο 2007 ως 2013. Επίσης, κατοχυρώσαμε την η κατανομή των χρηματοοικονομικών μέσων ανά δηλαδή αν πρόκειται για εγγυήσει, για δάνεια ή για τίτλους. Επίσης, ενοποίηση της διαχείρισης ανάμεσα στην Επιτροπή, δηλαδή και τις Εθνικές Συντονιστικές Αρχές και επίσης διάκριση, εξομάλυνση της διάκρισης ανάμεσα στις χώρες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και αυτές που δεν χρηματοδοτούνται το σε 7 κράτη-μέλη. Αναγνωρίζονται βέλτιστες πρακτικές από τη Γερμανία, από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την ε, Σλοβακία και την Εστονία. Δεν έχουμε ε, ικανοποιητικό δείγμα. με στόχο να διαμορφώσουμε μια σφαιρικότερη άποψη για αυτά τα μέσα, ανέλησε το ελληνικτικό συνέδριο ε, καλές ε, πρακτικές ε, προγραμμάτων με διεθνή καταξίωση, όπως ε, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης στη Γερμανία, δηλαδή τα γερμανικά ταμεία Marshall, όπως ονομάζονται, όπως είναι γνωστά. Επίσης, ένα πρόγραμμα στο Ισραήλ σε σχέση με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα αντίστοιχο αμερικανικό πρόγραμμα. Χρησιμοποιήσαμε ή μάλλον διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, συγκρίσιμα μέτρα ανάμεσα ε, σε όλα αυτά τα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη η διευκόλυνση ε, σύσταση νέων επιχειρήσεων, startup facility. Στη συνέχεια τα FEE e δάνεια ή τα δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ΣΜΕΚ, όλα αυτά τα μέσα έχουν παρεμφερεί σε στόχους όπως και τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή να, τονίσουν, να τονώσουν την ευημερία και να δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόληση και να βοηθήσουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει με τη χρήση νέων χρηματοοικονομικών μέσων. Υπάρχουν όμω και διαφορέ, ε, κυρίω ω προ του περιορισμού ε, τη κοινή διαχείριση ε, και ω προ του ευρύ εδαφικού χωροταξικού στόχου. Κρίνουμε ότι αυτή η σύγκριση που έγινε μα βοήθησε για τι μειονεκτού περιοχέ, ώστε να τυποποιήσουμε τι διαδικασίε και τον τρόπο αξιολόγηση. Επίσης, ε, αποτιμήσαμε τι επιπτώσει ε, των ε, κρατικών επιδοτήσεων με στόχο την άντληση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα και ο συντελεστή εμόχλευση που χρησιμοποιήθηκε υποδιαιρείται, μάλλον καλύπτει επίση και τα χρήματα που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα για την εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Μπορούμε να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα της έκθεσής μας σε τρεις βασικούς τομείς. Πρώτον, ε, η ποιότητα της αξιολόγησης των δανειακών αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από αυτή την πλευρά, για την προγραμματική περίοδο 2000 2006 δεν έγινε καμία τέτοια αποτίμηση. Η κατάσταση άλλαξε για την επόμενη περίοδο, 2007 2013 δηλαδή, όπου ε, παρά την απουσία νομικής τυπικής υποχρέωσης ε, ενθαρρύναμε την αξιολ. και χρηματοδοτήσαμε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την αξιολόγηση βάσει του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου κατόπιν ετήματος των κρατών μελών. Επίσης, ποσοτικοποιήσαμε την ανάγκη παρέμβασης του δημοσίου τομέα. Εκεί σημειώθηκε πρόοδος. Η ποιότητα αυτής της αξιολόγησης διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από κράτος σε κράτος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 οι αξιολογήσεις αυτές ε, έγιναν με ανεξάρτητο τρόπο, στα πλαίσια δηλαδή του επιχειρησιακού προγράμματος. Ε, δυστυχώς υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις και ως εκ τούτου δεν κατανεμήθηκαν με ικανοποιητικό ε, τρόπο τα κονδύλια, ανάχρημα το οικονομικό μέσα. Δεν έγινε επίσης ανεξάρτητη αναθεώρηση αυτή τη αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Σεπτέμβριο του 2011 εξέδωσε μία έκθεση όπου χαρακτηρίζει τις δανειακές ανάγκες ως εν μέρη την κάλυψη των δανειακών ανακών ω εν μέρη μη ικανοποιητική και ε, παραθέτει και κάποιου λόγους ε, που ενδεχομένως αιτιολογούν την κατάσταση. Ο δεύτερο τομέα ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΤΠΑ για την χρήση και υλοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Εδώ η βασική επίκριση που απευθύνει το ελεγκτικό συνέδριο συνδέεται με το ότι παρά την αυξανόμενη οικονομική ε, σημασία αυτών των μέσων, ε, ε, τα διορθωτικά ταμεία και οι σχετικοί κανονισμοί για το 2007 2013 δεν έλεβαν κατά το δέον υπόψη την, τις ιδιαιτερότητες του κάθε χρηματοοικονομικού μέσου. Ως αποτέλεσμα εφαρμόζονται αυτά τα μέσα χρησιμοποιώντας τη νομική βάση που όμως είχαμε αρχικά σχεδιάσει για τις επιδοτήσεις. Οπότε τα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης δεν προβλέπουν Βλέπουν επαρκή ε, διαχείριση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσεων. Ε, και ένα σημαντικό προσανατολισμό λάβαμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Φεβρουάριο του 2011, εν μέσω δηλαδή τη προγραμματική περίοδου και σίγουρα όχι εγκαίρω. Ε, επιπροσθέτως, λόγω ε, της μορφής που πήρε ο προσανατολισμός που μας προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή δεν είναι δεσμευτικός, ε, παρακολεί ε, τη δυνατότητα, το δυναμικό των χρηματοοικονομικών αυτών ε, ε, μέσων, δεν τα αφήνει να αναπτύσσουν αναπτύξουν πλήρω την οικονομική τους ε, ε, δύναμη. Θα ε, ναι, αναλύσω ακόμη βαθύτερα το θέμα. Το συνέδριο διαπίστωσε τέσσερις βασικές ατέλειες που, παρα, που παραμένουν παρά τι εξηγήσει και τον προσανατολισμό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, δεν υπάρχει επαρκή μόχλευση ούτε και διατάξεις σε σχέση με τη λειτουργία, βάση δηλαδή οικονομικού έτου ή όχι του Ταμείου έτσι μακροπρόθεσμα υποσκάπτονται ε, και δεν μεγιστοποιούνται τα ωφέλη των χρηματοοικονομικών αυτών ε, μέσων. Επίσης, ε, είναι δυνατόν μη αιτιολογούμενα κονδύλια να αποδοθούν, να καταλογιστούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Παραδείγματο χάρη, υπάρχει μια υπερμεγέθηση πρικοδότηση ενός ταμείου. Σας παραπέμπω σελίδα 25, πίνακα σε 2. Ε, στη συνέχεια υπάρχει δυνατότητα να προσφεύγουμε ανεφετιολογήσεως σε διακριτική μεταχείριση ως προς τον ιδιωτικό τομέα. Ε, ελοχεύουν οι κίνδυνοι ούτως ή άλλως με τα αμοιβαία κεφάλαια και με αυτές τις διατάξεις φέρει ολόκληρη την ευθύνη ο δημόσιος τομέας και η ρήτρα ε, αναδιάρθρωσης ε, δεν ε, καλύπτει τις απαιτήσει που θα έπρεπε για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, κυρίως προς το κεφάλαιο κίνησης. Σε σχέση τώρα με την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων υπάρχουν τα θέματα κοινή διαχείρισης, όπως σας είπα, το θέμα της, του χωροταξικού σχεδιασμού που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και επίσης η ανάγκη υιοθέτησης σε μια κρίσιμη μάζα, ούτως ώστε να είναι βιώσιμα αυτά τα προγράμματα ε, και να μην έχουμε τις, ε, ε, τις γενικές δαπάνες να υπεσκελίζουν την αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων. Χρειαζόμαστε ε, μεγαλύτερη διαφοροποίηση επίση, ούτω ώστε αποδέκτε να είναι ακόμη περισσότερε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, το συνέδριο ε, αξιολόγησε επίση την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών μέσων του ΕΤΠΑ για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ω προ την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Οι επιδόσει επηρεάστηκαν αρνητικά από ευρέω διαδεδομένε καθυστερήσει ω προ την χρήση αυτών των μέσων. Έτσι, το βασικό πλεονέκτημα αυτής της ε, αποπληρωτέας ε, βοήθειας ε, ακυρώνεται. Ε, δηλαδή δεν μπορέσαμε να ε, ανασυστήσουμε την πυρκοδότηση αυτών των ταμείων για την ε, περίοδο 2007 ως 2013. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τα ταμεία να υπερβούν την προγραμματική περίοδο. Γι' αυτό τον απλό λόγο. Επίσης θα πρέπει να καταγράψουμε τις κακές επιδόσεις του ΕΤΠΑ ως προς την άντληση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα για αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα εν συγκρίση με άλλα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, καλό θα ήταν να κάνουμε διάκριση αναταμία. Π.χ. τα ποσοστά μόχλευσης ε, ήταν υψηλότερα σε κάποια ταμεία. Επίσης είχαμε Ε, σημαντικές διαφορές στο ίδιο κράτος μέλος ε, σύν χρόνο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι ρυθμίσεις έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τις βασικές αδυναμίες που αναφέραμε. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε πως τα μελλοντικά μέσα θα συστήνονται μόνο μετά από εύρωστη αξιολόγηση του καινού χρηματοδότησης και βεβαίως η κατανομή των κονδυλίων θα συμφωνεί με αυτή την αξιολόγηση το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να προσαρμοστεί στη φύση και τα χαρακτηριστικά των ε, χρηματοδοτικών μέσων για να μην έχουμε τις ελλείψεις οποίες έχουμε. Εν τω μεταξύ ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει και ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός και μια πρόταση για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο μετά το 2013 είναι ήδη προτάσεις του νομοθέτη. Το δικαστήριο έχει ε, γνωμοδοτήσει και για τα δύο αυτά νομοθετήματα. Αυτά τα παρουσίασε οι συνάδελφοι ε, Φάζακας και Μπόστοκ ε, στην Επιτροπή σας. Ε, συνολικά θεωρούμε πως οι προτάσεις αυτές ως έχουν, αντιμετωπίζουν εν μέρη το πρόβλημα που μόλις ανέφερα. Το δικαστήριο συνιστά στα κράτη-μέλη ή δυνατόν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που υπάρχουν στο ΕΤΠΑ για να ενσωματωθούν όλα τα ε, συγχρηματοδόμενα προγράμματα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Π.χ. το έχει κάνει αυτό η Πορτογαλία με θετικά αποτελέσματα. Τα νομισματικά συστήματα και τα συστήματα ελέγχου επίσης θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως και να διαχωριστούν από τις καθαρές επιχορηγήσεις. Ένα ε, μικρός αριθμός δεκτών θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ Κομισιών και Εθνικών Αρχών οι σημαντικές έννοιες της μόχλευσης και της ανακύκλωσης των κονδυλίων θα πρέπει να οριστούν στον κανονισμό. Καλό θα ήταν για κάθε τύπο μέσου να οριστούν ελάχιστα ποσοστά μόχλευσης, ε, περίοδοι ανακύκλωσης και δεδομένα υπολογισμού αυτών των λόγων, αν και Βεβαίω δεν θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε κατά 100% με παρόμοια ιδιωτικά μέσα, Παρ' όλα αυτά, οι σαφείς στόχοι μας βοηθούν να επιτύχουμε τα αποτελέσματά μας. Η Κομισιόν επίσης θα πρέπει να δει την δυνατότητα να δίνει στα κράτη-μέλη έτοιμες λύσεις ε, χρηματοδοτικών ε, μέσων για μείωση του κόστους και γρηγορότερη εφαρμογή. Παραδείγματα αναφέρονται στην έκθεση τέλος, ε, εάν οι συστάσεις αυτές δεν μπορέσουν να εφαρμοστούν υπό το πλαίσιο του πολιτική συνοχής ε, καλούμε την Κομισιόν να ερευνήσει διαφορετικού τρόπους ε, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, θα ήθελα να τελειώσω, κυρίε και κύριοι, λαμβάνοντα υπόψη κάποια σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά από τον έλεγχο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χαιρόμαστε για το ότι η Κομισιόν δεν αδρανούσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου στην περίοδο αυτή η Κομισιόν έχει αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία ελέγχου των ε, μέσων χρηματοδότησης και έχει προχωρήσει σε μια τροπολογία των ε, κανονισμών με στόχο τα κράτη-μέλη να δίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των μέσων αυτών, αντιμετωπίζοντας έτσι τις συστάσεις που περιέχονται στην ετήσια εκθέση του συνεδρίου για το 2010. Επίσης, η Κομισιόν ε, έχει ε, συντάξει δύο σχετικά έγγραφα, το έγγραφο εργασίας ε, του προσωπικού για τα χρηματοδοτικά μέσα στην πολιτική συνοχή, στο οποίο θα παρουσιάσει ο κύριος Ντεφά στην Επιτροπή σας σήμερα και την έκθεση σύνθεση για την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων για το 2010 που καλύπτει κάποια γεννά πληροφόρηση για το πώς εφαρμόζονται αυτά τα μέσα σε ολόκληρη την Ένωση. Τέλος, ανέφερα ήδη την πρόταση για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ε, συνοχής μετά το 2013 και συγχαίρουμε την Κομισιόν και ελπίζω ειλικρινά όλα αυτά να συνεισφέρουν σε καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και Νόβακ. Νόακ πάρα πολύ σημαντική η έκθεσή σας για τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις ε, και ο κύριος Βαρόσο και ο κύριος ε, Ταγιάννη το τόνισαν είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας 99% των επιχειρήσεων έχουν κάτω από 250 εργαζόμενους άρα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής σας ευχαριστούμε για αυτά τα οποία μας είπε λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο είναι σημαντικό το ότι πρέπει να γίνει αυτή η λεπτομερής ε, συζήτηση, αλλά θα ήθελα τώρα, επειδή έχει προχωρήσει και ο χρόνος, αναφέρατε δύο έγγραφα, το έγγραφο εργασίας κομισιών ε, για, το, για τα μέσα χρηματοδότησης, ε, το οποίο θα μας, θα μας παρουσιάσει ο κύριος Ντέφα, τον οποίον καλωσορίζω, αλλά πρώτα απ' όλα θα γίνει μια σύντομη συζήτηση και σας παρακαλώ οι συνάδελφοι οι οποίοι ζήτησαν το λόγο, Φιέλνερ και Αγιάλα Σέντερ, να τοποθετηθούν σύντομα. Αλλά πρώτα απ' όλα, ε, εάν θέλει, ο κύριος Ριβελίνη, ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον ε, κύριο Νόατ για την ε, παρέμβασή του αλλά και για την ευγένεια που είχε. την προηγούμενη εβδομάδα συναντηθήκαμε, είχαμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων για να προετοιμάσουμε τη σημερινή συνεδρίαση. Στην ομιλία του μας παρουσίασε πολύ σαφώς τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου που έκανε το συνέδριο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα, ε, μέσα, ε, τα τεχνικά χρηματοπιστωτικά μέσα, χρηματοοικονομικά μέσα για την περίοδο 2006 Πολλά ακόμη πρέπει να εμπαθύνουμε, επειδή λοιπόν μου ζήτησαν να είμαι σύντομο, θα μιλήσω αποκλειστικά για τα θέματα που θεωρώ πως είναι τα πιο σημαντικά. Και καταληκτικά, αν με επιτρέψετε, θα σας πω και την προσωπική μου άποψη. Πρώτα απ' όλα, πολλά θα μπορούσα να πω για αυτά τα μη χιτάφ, ε, μας βοηθάνε πολύ αυτά τα μέσα για να ευνοήσουμε την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη κτλ. Αλλά δεν μπορούμε νομίζω να αγνοήσουμε το ότι υπάρχουν ε, αρκετές ε, ανεπάρκειες σε αυτά τα οποία διαπίστωσε στο συνέδριο. Πρώτα απ' όλα είναι εμφανές ότι υπάρχουν ε, κατάφορες ανεπάρκειες όσον αφορά το αποτέλεσμα μόχλευσης το, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιδιώκουμε και το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό, αν αναλύσουμε το σύνολο των στοιχείων, διαπιστώνουμε σαφώς ότι το μοχλευτικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ταμεία τίτλων, στα πλαίσια του ΕΤΠΑ, περνάμε από το 1 στο 2,75, δηλαδή κυμαίνονται μεταξύ 1 και έως 2,75. Και αν αναλύσουμε το, το αποτέλεσμα μόχλευσης ε, μέσω δανείων, περνάμε ότι διαπιστώνουμε ότι είμαστε μεταξύ 1 και 1,67. Είναι ακόμη δηλαδή πιο σοβαρή η κατάσταση. Και η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τρόπος χρηματοδότησης δεν υπολογίζεται σωστά. Δεν υπολογίζεται σωστά συγκεκριμένα το πολλαπλησιαστικό αποτέλεσμα. Η εθνική χρηματοδότηση πρέπει να είναι υποχρεωτική. Και πρέπει να υπολογίζεται σωστά το πολλαπλησιαστικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν όμω θετικά αποτελέσματα πολλαπλησιαστικά για τα μία εγγύσεων. Γιατί εκεί βλέπουμε ότι ε, πάει έω 4 το αποτέλεσμα αυτό. Θα ήθελα όμω συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε συγκεκριμένη επένδυση. Το ίδιο το συνέδριο δεν, μοιάζει να θεωρεί αξιόπιστα τα στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα ποσό 12 συνολικό. Θέλω λοιπόν μια γραπτή απάντηση και θα ήθελα στο πλαίσιο του δυνατού να έχουμε μια κατανομή αναταμίου και κράτος μέλος. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει νομίζω να μας απασχολήσει. Δεν έχουμε ανάλυση του κενού χρηματοδότησης, ιδιαίτερα για την περιοδο 2000-2006. Δεν βλέπω καμία ανάλυση του καινού χρηματοδότηση. Ούτε καν ζητήθηκε. Ενώ για την περίοδο 2007-2013, για την οποία ε, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, έχουν ζητήσει αξιολογήσει, για αυτή λοιπόν την περίοδο, με βάση τα στοιχεία του συνεδρίου, έχουμε 55 εκθέσει αξιολογήσει. Σημαντικό πολύ αυτό. Διότι νομίζω ότι οι αξιολογήσει του καινού χρηματοδότηση πρέπει να γίνονται. Οι αξιολογήσει αυτέ πρέπει να έχουν συγκεκριμένο στόχο, να μην αφορούν μόνο την χώρα που λαμβάνει, συνολικά δηλαδή, τη χρηματοδότηση, αλλά τι περιφέρειε τη χώρα αυτή. Οπωσδήποτε θα έχω τη δυνατότητα αυτά τα στοιχεία να τα αναφέρω στην έκθεσή μου, μόλι θα έχουμε αξιόπιστα στοιχεία για κάποιες μορφές συγκεκριμένες χρηματοδότηση, για κάποιες περιφέρειες της Ένωση θα πρέπει να ευνοηθούν σε σχέση με άλλες. Θεωρώ λοιπόν ότι τα μέσα χρησιμοποιούν κεφάλαιο υψηλού κινδύνου δεν είναι τα κατάλληλα και πρέπει να χρησιμοποιηθούν περιορισμένα. Πρέπει να ευνοήσουμε περισσότερο τα μέσα εγγύσεων στις πιο ευαίσθητες περιοχές. Για τις περιόδους που ανέφερα, δεν νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα μέσα και δεν νομίζω ότι είχαμε τις σωστές εκθέσεις οι αιτήσει εκθέσεις και τα άλλα μέσα που χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση δεν νομίζω ότι αποτιμούν σωστά την ειδική φύση αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων. Έχουμε στοιχεία που μας αποδεικνύουν ότι ορισμένε φορές η χρηματοδότηση δεν αξιοποιήθηκε για τον σκοπό για τον οποίο είχε κρεθεί Και αυτό αποτέλεσμα η Ανταλουσία. Λόγω αυτών των ανεπαρκειών που μας δημιουργούν ε, πολλές απορίες, θα θέλαμε τα χρηματοπιστωτικά αυτά μέσα να τα θεωρήσουμε αρνητικά. Θα υπήρχε αυτός ο πειρασμό. Όμως έχουν αξιόλογο δυναμικό για την Ευρώπη, αξιόλογε προοπτικέ, οπότε συστολικά η αποτίμησή μου παραμένει θετική. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην νομική και επιχειρηματική πλατφόρμα που χρησιμοποίησαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ίσως και εκείνη αντιλήφθηκε τις ανεπάρκειες, τις πολύ συγκεκριμένες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι δημιουργήσαμε χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν έχουν ένα συγκεκριμένο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο και άρα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός στο τίτλο 8 ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε μια σειρά από θέματα που υπάρχουν και που δημιουργούν νομικές ασάφειες και αβεβαιότητες. Θεωρώ ότι εάν το νομικό πλαίσιο που θα έχουμε στο μέλλον είναι αυτό στο οποίο στοχεύουμε, ιδιαίτερα στα πλαίσια του τίτλου 8 του σχεδίου δημοσιονομικού κανονισμού, δημοσιονομικού κανονισμού θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα όπω ακριβώ προβλέπει και το συνέδριο. Επίση, θα ήθελα να καλέσω το συνέδριο να μου πει, ενδεχομένω γραπτό, ποιο είναι το επιχειρησιακό κόστος και το κόστος διαχείρισης των ταμείων αυτών. Γιατί διαβάζοντας την έκθεση αυτή δεν είδα αυτά τα στοιχεία. Και στρέφομαι και προς την Επιτροπή και θα ήθελα λεπτομέρειες επιπλέον. Για παράδειγμα, πώς θα υπάρξει συνέπεια μεταξύ των κατεξοδότηση πράξεων και των επιχειρησιακών αποφάσεων. Ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί δράσης που έχουν στόχο να λάβουν υπόψη την ανακοίνωση που έγινε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο 662-2011. Τέλος, πιστεύω πως θα ήταν επίσης σκόπιμο να υπάρξει εναρμόνιση των μεθόδων εργασίας και ανάλυσης. Οι παράμετροι, οι δείκτες που χρησιμοποιεί το συνέδριο και η Επιτροπή διαφέρουν σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα ουσιαστικά στοιχεία. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνουν όλε οι αναγκαίε προσπάθειε για να εναρμονιστούν οι μέθοδοι εργασία. Νομίζω ότι είναι ουσιώδε. Επαναλαμβάνω. θέλω να μάθω ποια είναι τα ακριβή ποσά των χρηματοδοτήσεων που δίδονται και για κράτο μέλο και ανατύπω ταμείων. Και ευχαριστώ τον Δόκτορα Νόακ για την ευγένειά του και την έκθεση που μα παρουσίασε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ριβελίνη. Ο κύριος Φιέλνερ χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Τα μέσα αυτά διαχείρισης χρηματοδότησης ήταν κάτι το οποίο μας προκάλεσε πονοκεφάλους στη διαδικασία απαλλαγής και επιδεινώσατε αυτό το πονοκέφαλο γιατί όπως και η ίδια η Κομισιόν σωστά συμπέρανε πρόκειται για έργα υψηλού κινδύνου αλλά ε, σημαντικότερο το ότι δεν ε, έχουμε νομικά μέσα για να τα διαχειριστούμε και το είπατε αυτό σαφώς. Τούτου τελευταίο όμως πρέπει να πω και συμφωνώ με τον κύριο Ριβελίνη πως ε, θεωρώ πως υπάρχει κάποιος ρόλος που μπορούν να παίξουν αυτά τα μέσα αλλά πρέπει να είναι περιορισμένος καθορισμένος σωστά και να βασίζεται σε μία εκτενή αξιολόγηση του πότε ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν, αλλά έχω δύο ερωτήσεις έχοντας διαβάσει την παρουσίασή σας. Πρώτα απ' όλα βλέπω πως ε, τα μέσα αυτά χρηματοοικονομικής ε, τεχνικής ήταν κάτω από την λεγόμενη κρίσιμη μάζα, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν ε, πώς δίνει κίνητρα ο κανονισμός για να έχουμε μέσα τα οποία θα φτάσουν σε μια κρίσιμη μάζα, ειδικά μετά την ε, χρηματοδότηση αναπεριφέρεια. Ίσως θα μπορούσε το ελληνικό συνεδρίο να μας εξηγήσει κατόπιν. Στην ε, σελίδα 7, στο έγγραφο εργασίας της Κομισιόν, ε, υπάρχει μία παράγραφος ε, η οποία με εξέπληξε κάπως γιατί εκεί πέρα αναφέρεται πως η Κομισιόν ακόμα χρειάζεται εκθέσεις οι οποίες είναι εθελοντικές από πλευρά των κρατών μελών για να προετοιμάσει την αναφορά του 2011. Ξέρουμε πως αυτό ήταν πρόβλημα το 2010. Εδώ πέρα λέει πως ε, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα το 2011. Μα εγώ φανταζόμουν πως ο τροποποιημένος κανονισμός που ενέκρινε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πέρσι το Δεκέμβριο θα είχε λύσει το ζήτημα. Γιατί δεν ε, το αντιμετωπίσαμε τότε. Ε, ίσως θα μπορούσε να μας εξηγήσει η Κομισιόν. Αυτό ήταν πρόβλημα και το 2010, το ξέραμε πριν υιοθετήσουμε την νομοθεσία πέρσι το Δεκέμβρη, γιατί δεν το αντιμετωπίσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από πλευράς διαδικασίας να σας υπενθυμίσω πως η έκθεση Ριβελίνη ε, θα υποβληθεί 30 Μαΐου 2012 και θα υπάρχει δυνατότητα να την συζητήσουμε. Επειδή το ελεγκτικό συνέδριο ζήτησε η έκθεση αυτή πέρα από την παρουσίαση της ε, Κομισιόν, η οποία ούτως ή άλλως πρέπει να γίνει πριν τις 11.30 να συζητηθεί η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, παρακαλώ τους ε, συναδέλφους να περιοριστούν στην έκθεση αυτή για να έχουμε μετά χρόνο για τη συζήτηση και με τον κύριο Ντέφα. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ, μετά Γκρέσλε, Σταυρακάκης και η κυρία Βάνοβα. Παρακαλώ, κύριε Σέντερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Νόακ για την παρουσίασή του που ήταν τόσο διευκρινιστική και εκπαιδευτική γιατί προετοιμάζουμε τώρα τους κανονισμούς για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Είναι λοιπόν ένα από τα καινοτόμα στοιχεία αυτό, η χρήση αυτών των νέων μη μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για να αξιοποιήσουμε τον περιπολισμό της Ένωσης και να το συνδυάσουμε με το ειδικό κεφάλαιο. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί κάπου λέει ότι οι θετικές επιπτώσεις της χρήσης αυτών των μέσων για τις ΜΜΕ δεν ήταν όσο θα έπρεπε όσον αφορά τη συμβολή του ιδιωτικού κεφαλαίου από άλλου τύπου προγράμματα στα πλαίσια της Ένωσης για τις ΜΜΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί, γιατί δεν είναι συνηθισμένες οι ΜΜΕ σε αυτό το νέο μέσο, είναι πιο συνηθισμένες σε άλλο και ποια άλλα μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις ΜΜΕ. Ποια μέσα ήταν πιο ικανά να προσελκύσουν ιδιωτικό κεφάλαιο γιατί από τις μεταφορές και τον τουρισμό που ξέρω έχουμε μεγάλες δυσχέρειες τη στιγμή που προσπαθούμε να συνδυάσουμε δημόσιους πόρους με δυτικό κεφάλαιο. για την ε, μεγάλη διαφορά του κανονιστικού πλαισίου από αυτό, αυτό που θα, θα έπρεπε να είναι. Θα ήθελα να μου πει πού ακριβώς είναι τα σφάλματα που πρέπει να διορθώσει ο νέος κανονισμός. Γιατί λέτε ότι δεν είναι παρικές το κανονιστικό πλαίσιο. Το 2011, το Φεβρουάριο, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Θα ήθελα να μάθω εάν έχει λάβει αρκετές πρωτοβουλίες η Κομισιόν ή θεωρεί ότι χρειάζονται και άλλες. Επίσης, η συμβολή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά πόσο βοήθησε. Για κάποια μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε τώρα για τις μεταφορές, για παράδειγμα, η συμβολή και η τεχνογνωσία της ε, ΕΤΕ είναι πολύ σημαντική και κάποιων άλλων εκτελεστικών οργανισμών. Επαρκούν λοιπόν αυτοί οι φορείς χρειάζονται και άλλοι. Και τέλος, ο κύριος Νοάκ ανέφερε τη δυνατότητα ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν ε, αυτά τα μη ΤΑΦ από τις καθαρές επιδοτήσεις. Τι ακριβώς εννοεί. Αυτά τα μη ΤΑΦ για μεγάλα προγράμματα, μακροπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα, τι κάνουν. Ένα τμήμα είναι επιδοτήσεις και τα άλλα είναι δάνεια. Αυτός ο διαχωρισμός πρέπει να είναι μόνιμος, είναι κάτι το παροδικό. Και μιλάτε για πολύ διαφορετικές χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία. Όπω υπόθηκε, υπάρχουν επιχειρήσεις με λιγότερο από πέντε εργαζόμενους που για κάποια χώρα μπορεί να θεωρηθούν μικρές, σε άλλες μεσές, σε άλλε μεγάλες. Θα ήθελα να δω αν λοιπόν υπήρξαν προβλήματα και με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αγιάλα Σέντερ. Κυρία Γκρέτσλε, ευχαριστώ. Πράγματι σημαντική αυτή η έκθεση μια που ήσασταν κι εσείς έτσι είχατε λόγω τεχνική διάθεση. Να σας πω κι εγώ ένα παραμύθι που ξέρουμε ε, για τα νέα ρούχα του αυτοκράτορα. Δυστυχώς ο αυτοκράτορας είναι γυμνός. Όλα αυτά τα μέσα τα οποία υποτίθεται πως θα μας έβγαζαν από την οικονομική στενότητα δεν είναι διέξοδος. Εγώ βλέπω το διοικητικό κόστος και την ελάχιστη διαφάνεια γιατί Βλέπω πως ε, δεν έχει γίνει τίποτα ε, με βάση αυτά τα οποία μας ε, παρουσίασε το ελεγκτικό συνέδριο. Το πρώτο ερώτημα του ελεγκτικού, προς το ελεγκτικό συνέδριο είναι τι γίνεται με το διοικητικό κόστος. Δεύτερο προς την Κομισιόν. Η Γενική Διεύθυνση Έκθυνη είναι εδώ πέρα και πώς ερμηνεύει αυτή την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και τι συμπεράσματα βγάζει, γιατί αυτή η Γενική Διεύθυνση κατά την άποψή είναι υπεύθυνη για το ότι πιστεύουμε τόσο πολύ σε αυτά τα νέα ρούχα του αυτοκράτορα. Σας ευχαριστώ κύριε Σταυρακάκης. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Νόακ, ε, σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα έκθεση. Μοιάζει πάρα πολύ σημαντική για την πολιτική συνοχή, όμως το ελεγκτικό συνέδριο συνιστά να συμπεριληφθούν όλα τα μέσα του ΕΤΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ανά ε, χώρα. Σύσταση 7F. Δεν θεωρείται πως αυτό αντιβαίνει τη λογική της πολιτικής συνοχής η οποία παρεμβαίνει στο επίπεδο περιφέρειας. Οι ανάγκες ε, των διαφορετικών περιφερειών ε, μπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ και το να μπουν όλα σε ε, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν θα αυξήσει οπωσδήποτε την αποτελεσματικότητα των μέσων. Ευχαριστούμε κύριε Σταυρακάκη. Η κυρία Ιβάνοβα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, έλειπα σε μέρος της παρουσίασης λόγω της ψηφοφορίας στην Επιτροπή αλλά θα ήθελα να συγχαρώ το ελεκτικό συνέδριο. Εδώ στο Προεδρείο κάθομαι είναι σημαντική και επίκαιρη η έκθεση δεδομένης ε, της σημασίας των μέσων όχι μόνο λόγω της μόχλευσης αλλά και λόγω ακριβώ ακριβώς αυτής της ε, Ε, του ότι είναι κυλιόμενες ε, αυτές οι επιχορηγήσεις, δεν περιορίζονται σε ένα έτος, για να αντιληφθούμε την κρίσιμη σημασία τους για επιχειρήσεις, ε, ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάποιοι τομείς αναφέρθηκαν, εγώ θα αναφερθώ σε δύο μόνο. Μον έχουμε το κενό αυτό μεταξύ ζήτησης και διαθεσιμότητας των κονδυλίων και το δεύτερο σημαντικό ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε ε, επανειλημμένως όχι μόνο σήμερα η έλλειψη ξεκάθαρων δικτών και μέσων σύγκρισης είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αν δεν υπάρχει κάτι ε, για να συγκρίνουμε και το ερώτημά μου προς το ελεγκτικό συνέδριο είναι λέτε εδώ πέρα πως θα προτείνετε να εξεταστούν διαφορετικοί τρόποι στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με βάση αυτό το οποίο είπε και η κυρία Γιάλα Σάντερ ε, ποιο ρόλο βλέπετε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εδώ πέρα για να δούμε ακριβώς εναλλακτικούς τρόπους στήριξης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προς την Κομισιόν ένα ερώτημα. Ποια συγκεκριμένα μέτρα και βήματα θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις, ειδικά στην ανάλυση εξ άντε που πρέπει οπωσδήποτε να επιταχυνθεί. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, δεδομένου του ότι μέχρι τις 30 Μαΐου έχουμε χρόνο για να ασχοληθούμε με αυτή την έκθεση, σας παρακαλώ κύριε Νόακ συντομότατα εντός ε, τριών λεπτών να αναφερθείτε στα ζητήματα αυτά γιατί έχουμε και πολλές ερωτήσεις που απαιτήθηκαν ε, προς την Κομισιόν και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα απαντήσετε γραπτώς ή στις ε, επόμενες συζητήσεις. εντάξει. Σύντομα λοιπόν για αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και μέχρι τις 30 Μαΐου θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Κύριε Νόακ. Ναι, βεβαίως κύριε Πρόεδρε, αλλά να τονίσω πως το αντίστοιχο συνέβη. Εμένα μου ζήτησαν εάν ήμουν α, διατεθειμένος να απαντήσω τώρα κανονικά. Είναι άλλη διαδικασία και ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα να τονίσω πως δεν είναι τα πάντα σπρώμαυρα. Εάν χρησιμοποιήσει κάποιος ε, τα νέα μέσα, βεβαίως πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα υπόδειγμα και ένα πλαίσιο το οποίο θα λειτουργεί. Δηλαδή τα μέσα αυτά δεν είναι μόνο δάνεια, τα δάνεια τα δίνει κανείς και μετά του τα ξεπληρώνει, στη χειρότερη περίπτωση τα χάνει. Με τα μέσα αυτά τα χρηματοοικονομικά θέλουμε να επιτύχουμε κάτι παραπάνω. Οπότε χρειάζονται περισσότεροι και επαρκέστεροι κανονισμοί. Και άρα φτάνουμε σε ένα από τα ερωτήματα. Πράγματι, δεν μπορούμε σε όλα τα κρατημένα να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα. Παραδείγματο χάρη στα λιγότερο προχωρημένα και ανεπτυγμένα κράτη-μέλη είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε τα συνήθι μέσα τα δάνεια γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης τέτοιων ε, μέσων χρηματοοικονομικών γιατί αυτό σημαίνει πως χρειάζονται ενδιάμεση τράπεζες οι οποίες έχουν εμπειρία σε αυτόν τον τομέα οπότε πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση και άρα ερχόμαστε σε ένα άλλο ερώτημα στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μεγάλη ικανότητα και εντός της Κομισιόν και κυρίως εντός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν αυτά τα σύγχρονα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και συνεισέφεραν στην ε, διαχείρισή τους ε, νομίζω με τρόπο ιδιαίτερα έμπειρο. Ετέθη το ερώτημα το εάν συμφέρει αυτή η χρηματοδότηση. Εάν ξέρει κανείς τον κίνδυνο και έχει την αυτοπεποίθηση να διαχειριστεί αυτόν τον κίνδυνο, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά για να διαχειριστεί τον κίνδυνο χρειάζεται κανείς κανόνες και εμπειρία. Αυτά πάνε μαζί. Εάν μου επιτρέπετε, στις ε, περιπτώσεις που υπάρχει εντύπωση πως δεν υπάρχει εμπειρία, είναι καλύτερο να υπάρξουν επιχορηγήσεις, όπως κάναμε στο παρελθόν. Και να μην ε, αναζητούμε, παραδείγματος χάρη, ιδιωτικά κεφάλαια ε, για τις δημόσιες δαπάνες. Πράγματι, δεν υπάρχει αμφιβολία πως ε, τον θέλουμε να προσελκύσουμε δημόσια κονδύλια, με βάση τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του κάθε ευρώ, τότε τα ιδιωτικά κονδύλια δεν μπορεί να είναι κονδύλια των κρατών μελών, πρέπει να είναι ιδιωτικά, όντως. Και έρχομαι έτσι στο ερώτημα του γιατί δεν είναι σε κάθε περίπτωση δυνατόν να προσελκύσουμε ιδιωτικά κονδύλια. Μα αυτό είναι ζήτημα του ότι προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρο στις μικρομισές επιχειρήσεις. Δεν είναι κάθε επιχειρήση προσανατολισμένη προς το μέλλον ε, και προς τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Άρα ο ιδιωτικός τομέας εξετάζει κάθε φορά το επιχειρηματικό μοντέλο και συμμετέχει ή όχι. Παραδείγματος χάρη ε, αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι οι κατάλληλες για να ε, χρησιμοποιήσουμε πιο σύγχρονα μέσα χρηματοδότησης. Μου ζητήσετε πληροφορίες για το κόστος διαχείρισης. Σε ένα πρώτο σχέδιο τις έχουμε συμπεριλάβει και μπορούμε βεβαίως να σας δώσουμε τα στοιχεία ο κύριος Μούλτερ νομίζω τα ζήτησε. Οπωσδήποτε θα ε, σας δώσουμε τα στοιχεία των αμοιβών. Εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί οι αμοιβέ ε, κινούνται σε ε, μια ψαλίδα και είναι συγκρίσιμη νομίζω η διαχείριση τέτοιων ταμείων. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε μεγαλύτερες αμοιβές από τις άλλες περιπτώσεις κύριος Φιέλνερ ε, ρώτησε τι γίνεται με τις εκθέσεις. Να πω το εξής. Εάν δημιουργηθεί ένα ταμείο συμμετοχών και η Κομισιόν ή ο Ευρωπαίος φορολογούμενος είναι ο ιδιοκτήτης κατ' ουσίαν αυτού του ταμείου, ε, σε μια φυσιολογική εταιρεία υπάρχει ένα σύστημα αναφορών και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τα μία. αυτά πρέπει να δίνουν αναφορές ε, αναμήνα, τρίμηνο ή ετησίως. Εθελοντικά είναι μια ιδέα, αλλά νομίζω πως σύνηθες είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται να δίνουν αναφορά στον ιδιοκτήτη. Είναι νομίζω συνήθις πρακτική. Τελευταία ερώτηση. Ε, τον κύριο Σταυρακάκη. Ε, πρέπει να δείτε την κατάσταση στην περιφέρεια στην οποία θέλει κανείς να ε, ξοδέψει λεφτά και βέβαια ο τίτλος είναι η πολιτική την οποία θέλει να αναπτύξει. Και μετά βέβαια να αποφασίσουμε ποιο είναι το επαρκές μέσο για να χρησιμοποιηθεί εκεί πέρα. Και κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου π.χ. για να χρησιμοποιηθεί σε μια περιφέρεια. Δεν υπάρχουν τα μέσα για να γίνει κάτι τέτοιο, οπότε θα, θα αποτύχουμε. Εναλλακτικέ μέθοδοι, η τελευταία ερώτηση, νομίζω την ε, απάντησα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Ταμείο Επενδύσεων έχουν τις δυνατότητες να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε πως ε, όταν χρησιμοποιούμε νέα μέσα, χρησιμοποιούμε και νέους κανονισμού. και Πρέπει να έχουμε κατά νου πως όταν θέλουμε να επιτύχουμε περισσότερα με τα ίδια λεφτά υπάρχει περισσότερος κίνδυνος από το να δώσουμε απευθεία χρηματοδότηση. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε να μην ε, μακρηγόρησα. Ναι, ευχαριστούμε κύριε Νόακ για τις απαντήσεις αυτές ε, στις ερωτήσεις και θα ήθελα και εγώ να τονίσω το προσωπικό μου ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, το οποίο είναι μεγάλο, γι' αυτό συζητήσαμε λίγο περισσότερο. Και υπάρχουν τώρα και κάποιες ερωτήσεις προς την ε, Κομισιόν που πάνε πέρα από τα χρηματοοικονομικά μέσα. Το πώς γίνεται η ρύθμιση του τραπεζικού μας τομέα είναι ένα ερώτημα το οποίο συζητήθηκε και σε άλλες επιτροπές. Δεν θα πρέπει δηλαδή οι ρυθμίσεις αυτές και οι απαιτήσει ιδίων κεφαλαίων ε, να φτάσουν σε σημείο να μην επαρκέσει χρηματοδότηση και βλέπετε τι δυσκολίες έχουν οι μικρομισές επιχειρήσεις για να εξασφαλίσουν μικροχρηματοδότηση με χρηματοδότηση 5-10 ευρώ μπορεί να είναι αποφασιστική σημασία για την ε, ύπαρξη μιας επιχείρησης ή για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης αλλά βεβαίως ε, εάν ε, είναι σε ένα κεντρικό ταμείο με την ανάλογη αξιολόγηση ε, τότε όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε ίσως είναι πολύ υψηλό το κόστος διαχείρισης οπότε θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα μικρότερη προσφορά π.χ. Κομισιόν θα μπορούσε να το επιτύχει αυτό. Υπάρχουν λοιπόν κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Ντέφα ε, Υψηλέ προσδοκίες από την Κομισιόν για την μελλοντική ρύθμιση ε, αυτού του τομέα και τη βελτίωσή της. Και ευχαριστούμε ακόμη μια φορά κύριε Νόακ το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση αυτή για ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας απασχολεί. Και τώρα κύριε Ντίφα να έχετε τον λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε την ε, πρότασή σας για τα ειδικά μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής στην πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω και τα νέα μου καθήκοντα να μου επιτρέψουν να συνεχίσω την ε, καλή συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού όπως είχαμε καλή συνεργασία και όταν ήμουν εσωτερικός ελεγκτής. Θα ήθελα αν μου επιτρέπετε να μιλήσω αγγλικά, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο στο μέτρο το δυνατό. Το έγγραφο εργασία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά καλύπτει τρία ε, βασικά ζητήματα. Πρώτον, για ποιο λόγο είναι αυξανόμενο ο ρόλο των χρηματοοικονομικών μέσων στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή. Δεύτερον, ποια είναι τα βιώματά μα, οι εμπειρίε μα και ποια προβλήματα έχουμε εντοπίσει. Ε, επ' αυτού μας διαφώτισε ο κύριος Νόακ με την παρουσίαση των στοιχείων. Τον ευχαριστούμε και για την παρουσίαση και φυσικά για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Τρίτο σημείο και νομίζω ότι είναι και το πλέον βαρύνων. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής για να επιδιορθώσουμε αυτά τα προβλήματα. Θα ήθελα να σχολιάσω εν συντομία τα τρία αυτά ζητήματα. Λοιπόν, εντάχει για το πρώτο. Νομίζω η άποψή μας ε, απηχείται και στην παρέμβαση του εισηγητή εν μέρη, τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι πολύ σημαντικό τόσο ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε επιπρόσθετους πόρους για την ε, ανάπτυξη και για την απασχόληση. Ακριβώς δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Βιώνουμε μια κρίση, είναι περιορισμένα τα κρατικά κονδύλια και είναι καταπίγουσα η ανάγκη να ε, εξευρεθούν και άλλα κονδύλια για να μην επιστρέψω σε λεπτομέρειες, θα σας πω ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε μέσα από αυτά τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορεί να κινητοποιήσει και άλλα πολλά ευρώ για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και δεύτερον, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό, με την ομαδοποίηση των κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων, δεν ε, αντλούμε, απορροφούμε τα, μόνο τα κονδύλια, αλλά και την εμπειρία του ιδιωτικού τομέα. Πάρα πολύ σημαντικό και ισχυρότατο κίνητρο που θα ε, διασφαλίσει και την αηφορία αλλά και την ποιότητα των δράσεων. Αλλά προσοχή. Εδώ συζητούμε για τα χρηματοοικονομικά μέσα που ε, εφαρμόζονται στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Οπότε, χρηματοδοτούμε προγράμματα σε λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ, σε περιοχέ που αντιμετωπίζουν, εν πάση περιπτώσει, οικονομικέ δυσκολίε. Ε, για ε, στόχου δε που ε, δεν έχουν απαραίτητα βραχυπρόθεσμα ωφέλη, όμως μακροπρόθεσμα έχουν έναν υψηλότατο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και πάρα πολύ καλό δίκτυ κόστος ωφελίας, μακροπρόθεσμα. Ε, θα πρέπει να συνυπολογιστεί αυτό λοιπόν όταν χρησιμοποιείται μέτρα σύγκριση και εξετάζεται τους δείκτε επιδόσεων. Πιστεύω ότι δεν είναι πρόσφορο να αντιπαραβάλλουμε τις επιδόσεις των ταμείων στις μειονεκτούσες περιοχές με τις επιδόσεις τους σε ιδιαίτερα ανεπτυγμένες περιοχές. Παρόλα αυτά συμφωνώ ε, επί της σημασίας των δικτών επιδόσεων, όμως είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε μια προτιμησιακή μεταχείριση, ούτως ώστε να ε, ελκύσουμε ε, ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Όντως λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής, ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες και τις ειδικέ ανάγκες ε, κάθε περιοχής. Ε, περνώ στο δεύτερο θέμα, την εμπειρία μας. Αληθεύει ότι ήταν πολύ δύσκολη η ανηφόρα της εκμάθησης της όλης διαδικασίας. Η εφαρμογή των χρηματοοικονομικών μέσων σίγουρα ήταν πολύ δυσχερής. Όμως τώρα έχουμε μια σημαντική εμπειρία, θετική και αρνητική, Μέχρι τούτε λοιπόν σε τι αγγείται αυτή η εμπειρία μας. Ε, διαπιστώνουμε ε, αυξή σημαίνει χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων στην τωρινή περίοδο 0,5 από την ΕΤΕ, 0,7 από το ε, Ταμείο Επενδύσεων, όσο επιτοπλίστων χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την ανέπτυξη, για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για όλα τα ταμεία. Η ΕΤΕ και ε, το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Επενδύσεων έχουν εμπλακεί ενεργά και παρατηρήθηκε το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα επιπρόσθετη πόρη από εθνικά περιφερειακά κονδύλια από ιδιωτικού επενδυτέ ε, που όλα διαχετεύονται στα ταμεία αυτά, τα κεντρικά ταμεία που διαχειρίζονται με τη σειρά σου στα διαρθρωτικά ταμεία. Βεβαίως ε, δεν ισχυριζόμαστε ε, κάθε άλλο ότι είμαστε τέλειοι. Έχουμε εντοπίσει διάφορα προβλήματα και όπως προείπα ο κύριος Νόακ τα εξέθεσε με περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω ότι δεν είναι ικανοποιητική η ποιότητα των προγραμμάτων, η καθυστερήσει ω προ την εκταμείευση των κονδυλίων, η μη διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων, ε, χαμηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, μη ικανοποιητική μη μάζε, έλλειψη τεχνογνωσία ε, και κατευθυντηρίων γραμμών, υπερβολική πρικοδότηση, το ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι, αναπρόγραμμα. Ε, θα και όλοι ξέρουμε για ποιο λόγο, γιατί θέλουν κάποιοι να αποφύγουν τις δεσμεύσεις τους του N συν 2, N ε, συν 3, N συν 2 ε, και επίσης μη χρήση των ε, ε, ποιοτικών δικτών. Λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω με την εκτίμηση του ελεγκτικού συνεδρίου ότι η βασική αιτία του φαινομένου σχετίζεται με την σχέση ανάμεσα στην νομοθεσία και τι κατευθυντήριες γραμμές. Δεν μπήκαμε σε αρκετέ λεπτομέρειε. Ιδού το πρόβλημα. Τι έχουμε κάνει λοιπόν για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ε, ας αρχίσω με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Όπως ε, ανέφερε και ο κύριος ε, Νόακ, δεν έχουμε ε, αδρανήσει. Έχουμε αναλάβει δράσεις στους εξής τομείς. Ε, τεχνική αρρωγή και κατευθυντήριες γραμμές που διατίθεται πλέον στα κράτη-μέλη. Παραδείγματος χάρη, διευκρινίσαμε ότι για την εκαθάριση μόνο τα ποσά που έχουν ε, ληφθεί από τους τελικούς ε, αποδέκτες ε, είναι επιλέξιμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείτε να κρατάτε, να δεσμεύετε σε τα κονδύλια. Ως προς την ίδια τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων είχαμε καλύτερα αποτελέσματα σε ένα πρώτο στάδιο σε θελούσια βάση. Αντιλαμβάνομαι δε από αυτά που μας είπε ο κύριος Χέλνερ ότι δεν είστε ικανοποιημένοι προς το παρόν, όμως δεν σταματάμε εδώ. Όπως πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα έχουμε εισηγηθεί τροπολογίε για τον βασικό κανονισμό, οι οποίε θα προβλέπουν πλέον απαιτήσει λεπτομερεί απαιτήσει για υποβολή εκθέσεων. Όμως, ε, δεν έγιναν αποδεκτές όλες οι προτάσεις ε, που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θυμάστε ότι εσεί ε, ζητούσατε περισσότερα. Εμείς θελήσαμε να περιορίσουμε τις πληρωμέ σε δύο περιόδους επενδυτικών αναγκών. Το Συμβούλιο το απέρριψε αυτό. Υπήρξαμε και φιλόδοξοι, γι' αυτό το αναφέρω. Και καλό θα ήταν να ξέραμε νωρίτερα αυτά που βλέπουμε στην έκθεση. Επίσης, επιπρόσθετες ελεγκτικές ε, εργασίες ε, για να έχουμε ε, μεγαλύτερα εχέγγυα και να σφιγμομετρούμε την κατάσταση και φυσικά αρχίσαμε τις αξιολογήσεις. Αυτά για την τρέχουσα περίοδο. Για την επομένη... Έχουμε προτείνει ένα πολύ ολοκληρωμένο ε, νομικό πλαίσιο απαντώντας σε όλες τις ατέλειες που εντόπισε το ελεγκτικό συνέδριο. Οι προτάσεις για την αναθεώρηση του βασικού κανονισμού καλύπτουν ένα μεταξύ άλλων ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και βάσει των διατάξεων του κείμενου κανονισμού τονίζω ότι ένα από τα σημαντικά νέα στοιχεία είναι ότι ρίχνεται το βάρος στην ex αξιολόγηση που θα καλύψει ε, την ε, ε, μηνε χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών, την επαρκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, τη μόχλευση, την κρίσιμη μάζα, όλα αυτά τα ζητήματα δηλαδή που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των συζητήσεών μας. Επίσης, θα ε, ε, προτείνουμε μια ολόκληρη δέσμη λύσεων για την εφαρμογή. Ε, οργανισμοί επενδυτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης τυποποιημένα ετοιμοφόρετα, αν θέλετε, ε, μέσα και επίσης είναι προφανές ε, μέσα εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα. Για αυτά τα ετοιμοφόρετα, τα έτοιμα μέσα, ο στόχος είναι να επισπεύσουν την ταχύτητα εφαρμογής, ε, καλύπτοντας έτσι, απαντώντας έτσι σε μία από τις ανεπάρκειες που διαπιστώσαμε. Ω προ την χρηστή δημοσιονομική διαχείριση έχουμε κάνει και άλλε προτάσει και επανέρχομαι τώρα στην κάλυψη των επενδυτικών αναγκών για μια περίοδο που ανέχεται τουλάχιστον σε δύο χρόνια, αποφεύγοντα τα προβλήματα που ο κύριο ε, Νόκη, που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια τη συζήτηση, ε, τη υπερβολική δηλαδή ε, πρικοδότηση κάποιων μέσων, αποφεύγοντα επίση και τι διατότητε καταχρήσεων και παρατυπιών για τον κανόνα νήσιν 2. Σχετικά με τα τέλη, προτείνουμε επαναχρησιμοποίηση των πόρων για δεκαετή περίοδο και σαφείς δραστηριότητες υποβολής εκθέσεων παρακολούθησης και ελέγχου. Θα κλείσω, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει και απηχείται αυτό στι παρεμβάσει κάποιων συναδέλφων ότι παρόλα τα προβλήματα δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ε, το ισχυρότατο δυναμικό αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων στη χρήση του συγκεκριμένα στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή. Δηλαδή μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερα επενδύοντα σε λιγότερα. Αυτό ακριβώ δηλαδή που ε, χρειαζόμαστε ε, σε αυτή την περίοδο έλλειψη χρηματοδότηση. Έχουμε εντοπίσει δε προβλήματα που φυσικά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε και θα χρησιμοποιήσουμε και την γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου παρότι ε, σε κάποιους τομείς ε, θα διαφοροποιηθούμε κατά τι, ε, κυρίως ως προς τις ιδιαιτερότητες της πολιτικής συνοχής και ανάπτυξης της υπαίθρου. Θα ήθελα εντάχει να αναφερθώ στις παρατηρήσεις της κυρίας Γκρέσλε σε σχέση ε, με το Τζεάκφιν και την αντίδραση. Όταν διαβάζετε λοιπόν τι ε, απαντήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, να είστε σίγουροι ότι η Τζεάκφιν έχει εμπλακεί. Ε, και ότι οι απαντήσεις ε, που δίνουμε ε, προέρχονται από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Ήθελα να σας καθησυχάσω επ' αυτού. Λοιπόν, στο μέτρο του δυνατού στην ε, τρέχουσα περίοδο έχουμε επιδιορθώσει κάποια από αυτά τα προβλήματα και τώρα για την νέα περίοδο προτείνουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο που σε κάποιο βαθμό θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσει του ελεγκτικού συνδύου. Ε, προσοχή όμως, προς το παρόν είναι, ε, ε, πρόκειται για μία πρόταση και υπολογίζουμε στη δική σας υποστήριξη του συνομοθέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε αυτό το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τα, την χρηστή διαχείριση των δημοσιονομικών μέσων να μπορέσει να αποτυπωθεί στην νομοθεσία στο νομοθέτημα μόνο που τελικά ε, θα εγκριθεί. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά Ντέφα για την ε, ομιλία σας. Ελπίζω οι ερωτήσεις που τέθηκαν να μπορούν ε, τουλάχιστον εν μέρη να απαντηθούν. Ήταν περίπλοκες ερωτήσεις. Ελπίζω να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο. Ποιος θέλει το λόγο. Γκρέσλα και μετά και αν άλλη θέλει το λόγο ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Σπάνια ε, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε δουλευόμενοι, ε, να μάθουμε δουλεύοντα, συγγνώμη. Δηλαδή, ε, γι' αυτό ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ντέφα. Πραγματικά χαίρομαι που ήδη πέρασε αυτή η διαδικασία εκμάθησης τους, ε, που, στην οποία αναφερθήκατε και ελπίζω και η Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ να έμαθε όπως και εμείς. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε την υποστήριξη, είπατε, των νομοθετών. Η περιφερική Επιτροπή δεν υποστήριξε πολύ. Υπήρξε μια νέα εκπόνηση του κανονισμού αυτού και μετά εμείς δεν συμφωνήσαμε με τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Πιστεύω πως δεν θα πρέπει να συμβαίνει αυτό, ιδίως στο μέλλον για αυτούς τους μελλοντικούς κανονισμούς. Κύριε Ντέφα, μιλήσατε για αυτές τις κυλιόμενες ενισχύσεις για δεκαετή περίοδο. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αυτό για τον δημοσιονομικό κανονισμό, να δούμε πώς θα συνδυαστεί δηλαδή ο κανονισμός αυτός. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε και τη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα χρήματα, τα κυλιόμενα. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο και πληροφόρηση επαρκής δεν μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε το ύψος των απολειών. Πάντα υπάρχουν απώλειες, δεδομένο. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να μας κάνετε μια παρουσίαση για ποιου λόγου έχουν γίνει αυτέ οι παραλήψει που κοστίζουν χρήματα στο φορολογούμενο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο Γκάια. Ναι. Συζητάμε τακτικά στην Επιτροπή μας για τα χρηματοοικονομικά μέσα και νομίζω πως υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η μία λέει ναι, υπάρχει αρκετό δυναμικό να το εκμεταλλευτούμε. Ίσως ε, και η μόχλευση να μην είναι το τέλος αυτής της ε, διαδικασίας. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ περιθώριο βελτίωσης ε, και ακόμα δεν έχει εξαντληθεί νομίζω αυτή η διαδικασία εκμάθησης. Η άλλη σχολή σκέψης λέει πως ε, όσο δεν έχουν ρυθμιστεί και δοκιμαστεί τα μέσα αυτά και δεν υπάρχουν εγγυήσει για τη λειτουργία τους, καλύτερα είναι να μείνουμε μακριά. Εγώ είμαι στην πρώτη σχολή σκέψης. Θεωρώ πως ε, υπάρχει αρκετέ, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες στα μέσα αυτά χρηματοδότησης, αλλά βεβαίω αν ε, χρησιμοποιηθούν όπως μας είπε το ελεγκτικό συνέδριο τότε φοβάμαι πως ε, τα μέσα αυτά χάνουν την ελκυστικότητά τους πριν εξαντλήσουν ε, ολόκληρε, όλες τις δυνατότητές τους. Γιατί έριξα μια ματιά στις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και με χαροποιούν κάπως τα πράγματα τα οποία αναφέρονται εκεί πέρα, αλλά τι κάνουμε, ξεκινάμε εδώ πέρα μια πορεία με ένα πλοίο, εάν θέλετε, και μετά διαπιστώνουμε στη μέση της θάλασσας ε, πως ε, δεν είναι ε, το πλοίο αρκετά στεγανό, το πιδάλιο δεν λειτουργεί καλά ε, και ο καπετάνιος δεν πάει πολύ καλά. Μπορεί να ανακαλύψουμε και νέα γη παρόλα αυτά. Δεν ξέρω αν έτσι θα τα κατάφερνε ο Κολόμβος. Σε πάση περιπτώσει είναι ένα μεγάλο πείραμα. Θα δούμε τι θα γίνει και με την απαλλαγή του επομένου έτους της ε, Κομισιόν. Η κυρία Γκρέσλε μας είπε πως ε, με το Συμβούλιο δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι διαπραγματεύσεις ε, για το ζήτημα αυτό. Πώς θέλουμε λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε στη μόχλευση αυτή όταν επιμένει το Συμβούλιο πως οτιδήποτε επιστρέφει σε αυτά τα κυλιόμενα κονδύλια θα πρέπει να επιστρέφεται στα κράτη-μέλη. Εάν παραμείνουν σε αυτή τη θέση ε, μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό το μέσο εντελώ. Αλλά πιθανώ και το Συμβούλιο κάπου βεβαίως ε, στις Βρυξέλλες λειτουργεί και δεν ξέρει αριστερά του τι πει η δεξιά του. Αλλά Οι συνάδελφοι στις ε, αρμόδιες επιτροπές νομίζω πως ε, δεν ε, σκέφτονται ε, οπωσδήποτε το τι γίνεται σε άλλες επιτροπές θα μπορούσαν ίσως να τα δουν και να τα μεταφέρουν οπωσδήποτε στις πρωτεύουσές τους και να δουν μήπως ε, κάποιοι στο πλοίο το οποίο προανέφερα προσπαθούν να βουλώσουν τρύπες και κάποιοι άλλοι ανοίγουν νέες τρύπες στα ύφαλα. Αλλά το ερώτημα κύριε Ντέφα είναι εσείς θεωρείτε πως σας στηρίζουν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο σε αυτά τα οποία λέτε και σβήνει το μικρόφωνο του κύριου Γκάιερ. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο με ακούσατε, αλλά το ερώτημά μου προς τον κύριο Γενικό Διευθυντή ήταν το εξής. Έχετε την εντύπωση πως τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο σας βοηθούν στην προσπάθειά σας να κατευθύνετε αυτό το πλοίο στη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Γκάιερ. Ε, με συγχωρείτε κατά λάθος πάτησα το κουμπί σας. Λοιπόν, τελευταίος ο κύριος Μιλντερ να πω κάτι. Όλοι βεβαίως ε, χαίρονται πάρα πολύ για αυτά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα γιατί μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα με τα ίδια κονδύλια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εγγυήσεις δανείων κτλ. Υπάρχει κάποια εμπειρία τώρα, είδαμε κάποιες ελλείψεις ε, στο σύστημα και οπωσδήποτε θα αντιμετωπιστούν, αλλά αυτό το οποίο είναι πιο ενδιαφέρον για μένα είναι τι πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είχαμε. Και θα ήθελα πολύ περισσότερες πληροφορίε για τις μορφές που χρησιμοποιήθηκαν και ποια είναι η πιο επιτυχής. Με το νέο έτσι, πολυετές πλαίσιο να μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ των διαφόρων μέσων. Είναι ήδη σε θέση η Κομισιόν να κάνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Κύριε Μίλτερ, περνάμε λοιπόν στον τελευταίο γύρο απαντήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για τις ε, παρατηρήσεις της ε, κυρίας Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και για την αυτοκριτική ε, την οποία κάνατε και ελπίζω να μας στηρίξετε για τις νέες προτάσεις για το 2014-2020 με το πρόβλημα των ζημιών αναφέρατε θίξατε ένα σημαντικό ζήτημα και νομίζω πως ε, σήμερα δεν υπάρχει χρόνος ε, να το εξαντλήσουμε. Απλά ξέρετε πως ε, στα γερμανικά τι λεγόμενες επιχορηγήσεις είναι απώλειες. Τη στιγμή που το δίνετε δηλαδή πάνε τα λεφτά, χάθηκαν με τα ε, χρηματοοικονομικά αυτά μέσα υπάρχει τουλάχιστον η προοπτική να ξαναχρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα. Ναι, δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Εντάξει, μπορεί να υπάρξουν και ζημίες, αλλά ξέρετε, ο λογαριασμός θα βγει στο τέλος. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιες είναι όντως οι ζημίες. Δηλαδή πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε για ζημίες. Ε, να συγκρίνουμε και με την ε, εναλλακτική που υπήρχε. Που ήταν όπως σας είπα εξ αρχή χαμένες οι επιδοτήσεις. Ο κύριος Γκάιερ ε, αναφέρθηκε και οπωσδήποτε εμείς και εγώ το γνωρίζω πως έχετε και προσωπικό ενδιαφέρον και ως εισηγητής της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού για τα ζητήματα αυτά. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι πως ε, στη διάρκεια του έτους θα έχουμε καλύτερα δεδομένα, θα μπορούμε να δώσουμε καλύτερη αναφορά γιατί έχει αλλάξει και ο κανονισμός και τα κράτη-μέλη θα μας στείλουν τις ανάλογες ε, πληροφορίες. Οπότε θα έχουμε καλύτερες ε, πληροφορίες. Όπως είπα, κάνουμε επιπρόσθετους ε, ελέγχους και ε, θα καταλήξουμε σε μία αξιολόγηση. Οπότε και το ενδιαφέρον το ιδιαίτερο που επιδεικνύετε εσείς, οπωσδήποτε ε, το συμμεριζόμαστε κι εμείς και θα έχουμε καλύτερες πληροφορίες και ανάλυση. Όσον αφορά την στήριξη τώρα στο Συμβούλιο, δεν θα ήθελα να πω τίποτα. Να πω μόνο το εξής. Είναι σημαντικό πως όλοι πρέπει να δουν πως χρειαζόμαστε καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για αποτελεσματικότερα χρηματοοικονομικά μέσα στο μέλλον. Κύριε Μέλντερ, για πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ήδη ο ορισμός ε, την ε, παρονομαστής ε, και τι ε, διαιρέτης ε, μιλάμε για τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά μόνο, όλα τα δημόσια κονδύλια. Είναι δύσκολο επίσης να συγκρίνουμε εγγυήσει με δάνεια. ή με άλλα μέσα. Αλλά ελπίζω μέσω της, ε, των επιπρόσθετων ε, πληροφοριών και της αξιολόγησης να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να είμαστε σε θέση να κάνουμε σωστές ε, συγκρίσεις και να σας ενημερώσουμε στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Ντέφα για την ακρίβεια των απαντήσεών σας, την ε, δυσδυτικότητα, αλλά και για τις ε, λογοτεχνικές αναφορές. Ακούσαμε για τα για Χέσε, ακούσαμε για τα νέα ρούχα του αυτοκράτορα και ακούσαμε για τον Κολόμβο. Στον Κολόμβο δώσανε χρήματα για να πάει προς τις Ινδίες αλλά με καινοτόμο τρόπο ανακάλυψε κάτι άλλο που ήταν επίσης πολύ πολύτιμο. Καλό λοιπόν είναι εάν τα χρήματα που δίδουμε για κάτι ε, μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε κάτι άλλο θα μπορούσε να ήταν αυτό πολύ καινοτόμο. Βεβαίως μπορεί να ανακαλύψουμε κάτι άλλο από αυτό που ξεκινήσαμε να βρούμε αλλά εάν είναι χρήσιμο είναι θετικό το αποτέλεσμα. Το δίνει η γαρή μοίρα και το μέλλον αόρατο. Θα εξακολουθήσει να μα απασχολεί πολύ το θέμα αυτό. Αλλά βλέπετε, κυρία Γκρέσσα, έχει μια συμπληρωματική ερώτηση. Εάν θεωρήσουμε ότι όλα αυτά είναι πρόγραμμα κατάρτιση και υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα έπρεπε να έχει άλλη θέση στον προπολογισμό. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, βεβαίω. Βεβαίω. Αυτό θα βοηθήσει τον κύριο Γκάερ που πάντα ε, θέλει να ανακαλύψει νέα πράγματα. Εμείς ως υπεύθυνοι για τον έλεγχο του προπολογισμού πιστεύω ότι πρέπει να εξετάζουμε κατά πόσον αξιοποιούνται σωστά τα χρήματα, να μειώσουμε τις απώλειες και ελπίζουμε κύριε Ντέφα ο κανονισμό στο μέλλον να λειτουργήσει καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ που ήρθατε και απαντήσατε στι ερωτήσει μα. Κλείνουμε αυτό το θέμα τη μέρη διάταξη και επειδή έχει περάσει η ώρα θα σας πρότεινα τη συζήτηση για τη σημαντική επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην IT να την αναβάλουμε για την Δευτέρα. Μετά τις ψηφοφορίες θα έχουμε πιστεύω την επόμενη Δευτέρα αρκετό χρόνο. Για τα θα το κάνουμε κάπως βεβαιασμένα. Αν συμφωνείτε θα κλείσω την ε, δημόσια συνεδρίαση στο σημείο αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 26 Φεβρουαρίου και παρακαλώ να αποχωρήσουν όσοι δεν ε, ε, διατηρούν δικαίωμα παραμονής για να αρχίσει η